Uh, um, uh, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά δεν ήξερα ότι πρέπει να αντικαταστήσω τον ε, πρόεδρό μας, Ρομπέρτο Γουαλτιέρη, που θα έρθει σύντομα. Καταρχάς, καλώς ορίζουμε τα μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων από 15 κράτη-μέλη που είναι εδώ μαζί με τους συνεργάτες τους. Έχουμε, 10, έχουμε 56 συνολικά συμμετέχοντες από Εθνικά Κοινοβούλια για αυτή την ανταλλαγή απόψεων με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κύκλο του 2018 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Καλώς ήρθατε. Το σπίτι μας είναι και το σπίτι σας παρά το ότι μπορεί ορισμένες φορές να έχουμε κάποιες ε, έντονες συζητήσεις για να δούμε ποιος πρέπει να κάνει τι, αλλά πιστεύω ότι το βασικό είναι να συνεργαζόμεθα για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Είναι κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Εξαμένου του 2018 γιατί το Συμβούλιο πριν το καλοκαίρι υιοθέτησε τις συστάσεις του στα πλαίσια των αναχώρα εκθέσεων που θα εφαρμοστούν τώρα στο σχέδιο προπολογισμού που συζητάτε, στα σχέδια προπολογισμού που συζητάτε στα κοινοβούλια σας. Και επειδή η απόφαση που θα λάβει κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της έγκρισης των, σχεδίων, των νομοσχεδίων προϋπολογισμών μπορεί να έχουν επιπτώσεις σε άλλα νομοθετήματα είναι πολύ βασικό να συζητήσουμε μαζί τα πορίσματα από τον κύκλο 2018 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, η στάνταρ διαδικασία θα είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2018. Είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης, ε, αλλά δεν είναι απλή ολοκλήρωση. Ο συγκεκριτής ο κύριος Μαυρίδης είναι μαζί μας και στόχος μας επίσης είναι να συμβάλλουμε στη συζήτηση πριν εγκριθεί τυπικά η έκθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο 2018 πριν και αυτοί δημοσιοποιήσουν την τελευταία ετήσια έκθεση ε, οικονομικής ανάπτυξης που είναι θέμα επίσης κοινού ενδιαφέροντος. Εγώ απλώς θα φροντίσω για τα τυπικά και τα μαθαίνω πώς να τα φροντίζω αυτά όπως είναι τα καθήκοντα του Προέδρου όπως ε, ασκώ τα, τα καθήκοντα έχουμε 22 γλώσσες ε, σήμερα ευχαριστούμε τους διερμηνείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις κίτρινες κάρτες ε, για να ζητάτε το λόγο ε, δεν ξέρω αν στα εθνικά κοινοβούλια χρησιμοποιείτε κίτρινες κάρτες ε, για άλλα θέματα, αλλά εδώ θα είναι για να ζητήσετε το λόγο. Όποιο μέλος Εθνικού ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλει να μιλήσει, θα πρέπει να συμπληρώσει αυτή, αυτό το έντυπο που ήδη διανύμεται. Θα, διανέμεται. Ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαυρίδη να παρουσιάσει την έκθεσή του για να ξεκινήσει τη συζήτηση και κατόπιν θα δώσω το λόγο στους κοιόδης συζητητές εφόσον θέλουν το λόγο και κατόπιν θα δώσω το λόγο και ας πούμε σε δύο μέλη εθνικών κοινοβουλίων και μετά σε έναν ευρωβουλευτή, ένα λάξ, για να μπορέσουν όμως όλοι να πάρουν το λόγο. Ο χρόνος ομιλίας που θα έχετε θα είναι τρία λεπτά, όχι για τον εισηγητή. Ο εισηγητής μπορεί να πάρει λίγο περισσότερο χρόνο. Αλλά αν μιλήσει μισή ώρα σίγουρα θα τον διακόψω. Ευχαριστώ πολύ. Και να ξεκινήσουμε αμέσως με τον κύριο Κώστα Μαυρίδη. Ευχαριστώ κύριε Περβάους Μπερές που ασκείται καθήκοντα Προέδρου και εγώ θέλω να καλωσορίσω τα 20 μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων και τους 15, τις 15 αντιπροσωπείες κρατών μελών. Σας παρακαλώ να ε, βάλετε τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω ελληνικά. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. της αντιπροσωπείας των κρατών μελών. Η παρουσία σας και οι παρεμβάσεις σας είναι καθοριστικές στη σημερινή συζήτηση. Άλλωστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε εθαρρύνει τέτοιου είδους συζητήσεις και θεωρούμε προσωπικά και ως πολιτική ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών ότι αυτός ο διάλογος πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Ξεκαθαρίζω ότι η σημερινή μου πρωτολογία θα είναι επικριτική. Ωστόσο αναγνωρίζουμε και τη συνδρομή και συνεισφορά της Επιτροπής και των άλλων πολιτικών ομάδων σε όσους πιστεύουμε στο ευρωπαϊκό όραμα και στο ευρωπαϊκό εχείρημα. Η κριτική γίνεται γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε και να οικοδομήσουμε περισσότερο το κοινό μας μέλλον για να έχει μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι γιατί θέλουμε να το διαλύσουμε. Ξεκινώ λοιπόν λέγοντας ότι δεν μπορούσε να ήταν πιο επίκαιρη η σημερινή συζήτηση σε αυτή την έκθεση των ευρωπαϊκών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ. Κυρίως για τρεις λόγους. Αυτή η συζήτηση λαμβάνει χώρα λίγο πριν τη δημοσιοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης με τις οικονομικές και δημοσιονομικές προτεραιότητες για την επόμενη χρονιά. Δεύτερον, φυσικά επίκαιρο είναι και η συζήτηση για το τι συμβαίνει στην Ιταλία και τις σχέσεις της στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Θα επανέλθω σε αυτό. Τρίτον, να δηλώσουμε ότι βρισκόμαστε μόλις 7 μήνες πριν από τις ευρωεκλογέ. Για να έχει λοιπόν μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες να πιστέψουν στο μέλλον αυτής της Ένωσης. Πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινεί και να ενεργούμε αποφασιστικά, έχοντας πάντοτε ως οδηγό τις αξίες και τις αρχές μας, στις οποίες θεμελιώσαμε την Ένωση. Ομολογώ ότι άλλο πολλές φορές υποδεικνύουν οι δεσμευτικές μας αρχές και αξίες και άλλο κάποια φορά οι πολιτικές που ακολουθούμε. Και αυτό δυστυχώς τροφοδοτεί τον ευρωσκεπτικισμό και βάζει σε κίνδυνο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνω λοιπόν σε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Ολοκλήρωση της ΟΝΕ σε σχέση πάντα και με το τι συμβαίνει στην Ιταλία. Για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης απαιτείται ισχυρή πολιτική δέσμευση, αποτελεσματική διακυβέρνηση με βάση την κοινοτική μέθοδο και δημοκρατική λογοδοσία. Θα πρέπει επίσης να γίνεται καλύτερη χρήση των διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων. Τονίζω όμως ότι απαιτείται σωστή ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης. Αυτό είναι καθοριστικό για όσους πιστεύουμε και στα δύο. Μάλιστα, χαίρομαι καμιά φορά γιατί όσοι πιστεύουν στην αυτορύθμιση των αγορών 100% θυμούνται την εποπτεία και τη ρύθμιση δυστυχώς λίγο πριν την κρίση. Αυτό είναι μεν ευχάριστο, αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματικό, γιατί αν το σκεφτόμασταν εκ των προτέρων, πιθανώς να αποφεύγαμε κάποια από τα κακά που επισυμβαίνουν. Και με αυτό στο μυαλό θα είμαι πολύ πιο συγκεκριμένο σε ένα άλλο θέμα. Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχω πολύ έντονη άποψη, γιατί το έζησα εξ αρχής μέχρι σήμερα. Να θυμίσω λοιπόν ότι συμφωνήθηκε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση με τρεις πυλώνες. Δεν θέλω να μπω στη συζήτηση ποιο από τους τρεις πυλώνες συνέφερε σε ποιο κράτος μέλος. Συμφωνήσαμε μεταξύ μας ως ισότιμοι Ευρωπαίοι εταίροι σε τρεις πυλώνες. Εφαρμόσαμε τους δύο πρώτους και όμως γνωρίζουμε ότι ο τρίτος πυλώνας που είναι η πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων δεν εκπληρώνεται, δεν εφαρμόζεται, γιατί συγκεκριμένα κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτό λειτουργεί ενάντια στη δική τους εθνική ατζέντα. Και τονίζω ότι δεν είναι μόνο λόγοι οικονομικοί, είναι λόγοι και νομικοί και προπάντων ηθικοί μεταξύ μας. Συμφωνήσαμε τους τρεις πυλώνες και θα πρέπει να το εφαρμόσουμε και να μην βρίσκουμε προσχήματα για να το καθυστερούμε. Διότι κάθε μέρα που περνά οι αγορές μας δείχνουν ότι ελοχεύει και ένας νέος κίνδυνος με το να καθυστερούμε. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης αναφέρω ένα άλλο τεράστιο θέμα που αφορά τις αθέμητες πρακτικές και αθέμητες αθέμητους όρους, ιδιαίτερα σε καταναλωτικές συμβάσεις των τραπεζών. Μπορώ να αναφέρω πολλά παραδείγματα κρατών μελών, ξεκινώντας από το δικό μου, την Κύπρο, όπου υπήρξε μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις καταχρηστικές πρακτικές και του τραπεζικού τομέα η αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι απαραίτητη. Μεταξύ άλλων γιατί συμβάλλει και στον δίκαιο ανταγωνισμό. Ευρωπαϊκό εξάμεινο. Υπάρχει έλλειψη εφαρμογής των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων και εδώ χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μαθαίνοντας από τις μέχρι τώρα εμπειρίες μας, πιστεύουμε ότι υπάρχει έλλειψη εθνικής συμμετοχής στη διαμόρφωση και εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα και υποστηρίζουμε την αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με την ενσωμάτωση και νέων δικτών που θα αφορούν τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα. Είναι σημαντικό να θυμίσουμε εδώ τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενσωματώσει την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και με την διάσταση που απουσιάζει από τις συστάσεις αναχώρα για το 2018. Ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο είναι οι 20 βασικές αρχές και τα δικαιώματα που στηρίζουν τη δίκαιη και εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας. Αυτά ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Σκοπός μας είναι η επίτευξη καλύτερων συνθηκών ζωής και εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το πιστεύουμε, πρέπει να προτείνουμε πολιτικές και να τις στηρίξουμε. Άλλο θέμα. Ευελιξία κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας. Εξαιρετικά κρίσιμο και επίκαιρο. Θεωρούμε πολύ σημαντικό την ύπαρξη ευελιξίας κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως αυτό προτάθηκε και από την Επιτροπή το 2015 και θεωρούμε ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία για την τόνωση των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Υποστηρίζουμε στεναρά τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τη θέσπιση ενός συνολικού δημοσιονομικού προσανατολισμού της ζώνης του ευρώ. Σε αυτό θα περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, ο Υπουργός Οικονομικών και πολλά άλλα τέτοια θέματα. Τέλος, στο ίδιο θέμα, η ανάπτυξη νέων δημοσιονομικών εργαλείων με σκοπό τη σταθερότητα και την πραγματική σύγκληση των οικονομιών στη ζώνη του ευρώ. Και φυσικά η καταπολέμηση των κοινωνικών και οικονομικών αποκλήσεων. Να αναφέρω εδώ για παράδειγμα όχι μόνο την καταπολέμηση του εξτρεμισμού, αλλά την ανεργία, το brain drain, ιδίω από τον Ευρωπαϊκό Νότο και αλλού, όπου οι νέοι με τους νέους έχουμε το φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης. Απαιτείται λοιπόν αύξηση των πραγματικών μισθών, αφού είναι δεδομένο ότι είχαμε κατώτερη αύξηση στους μισθούς από ότι η παραγωγικότητα. Τέλος, ένα άλλο εργαλείο που ορίμασε ο καιρός, ένα λεπτό, just a minute, ρύθμιση ενός μηχανισμού για τον κατώτατο μισθό, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες του κράτους μέλους. Επιλεκτικά και μόνο αναφέρω τη σημαντικότητα των ταμείων συνοχής και ότι είναι απαραίτητο και θεωρούμε απαράδεκτες τις προτινόμενες περικοπές από την πολιτική συνοχής όπως προβλέπονται από την Επιτροπή. Και τέλος, επενδύσεις. Χρειάζεται ιδιαίτερη έμφαση, αναφέρω το πρόγραμμα Invest EU και τέλος Dear colleague, can you give the good example? I'm finishing up in 10 seconds. Just one sentence. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παιδεία. Δεν πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την παιδεία ως μοναδικό προσωρινό κόστος, αλλά με όλα τα πολλαπλασιαστικά εφέλη. Και τώρα είμαι έτοιμος να ακούσω τις δικές σας απόψεις σε αυτή τη συζήτηση που ξεκινάμε. Thank you, for your patience. Λοιπόν, Κοιτάξτε, ευχαριστούμε την Περβάνση για την υπομονή της, αλλά είναι για του φιλοξενούμενου μα υπομονή που θέλουν να μιλήσουν. Επιθυμούν διακαώ να μιλήσω γαλλικά. Να, να αλλάξω του κανόνε. Θα δώσω το λόγο εναλλακτικά σε σκιώδει εισηγητέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά σε δύο μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων. Με τη σειρά. ΕΛΚ. Για το Ευρωκοινοβούλιο. Πρώτη παρέμβαση. Τόμ. Βάντερ και μετά, ας ετοιμάζεται για την Ιταλία, ο Αλμπέρτο Ριμπόλα από την Έγκα του Βόρα. Τόμ, για τρία λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφοι των Εθνικών Κοινοβουλίων, με τα χαρά σα βλέπω εδώ και βλέπω ότι έχετε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμένου. Εγώ είμαι σκιώδη ηγητή για την ομάδα του ΕΛΚ όσον αφορά την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών Ζητημάτων για την οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Ας πούμε λοιπόν, ε, συνεχίζω πάνω σε αυτά που μας είπε και ο κύριος Μαυρίδης. Όπως γνωρίζετε κάθε χρόνο δημοσιεύονται συγκεκριμένες εκθέσεις αναχώρα που δεν είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Αν δεν θέλουν οι χώρες μπορούν και να μην συμμορφωθούν ταυτόχρονα, όμως βλέπουμε ότι η εφαρμογή των συστάσεων ε, πόρα απέχει από το Για το 2011-2017 παραδείγματο χάρη είμαστε στο 9% από την πλήρη εφαρμογή των διαφόρων συστάσεων. Ε, δύο είναι επιλογές ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και μπορούμε να διαπραγματευτούμε κάθε ομάδα μπορεί να παρουσιάσει ευχολόγιο, μπορεί να γίνουν συζητήσεις και ίσως μπορούν ε, να δούνε τι μπορεί να ενταχθεί ή να μην ενταχθεί στο ευρωπαϊκό εξαμήνο. Ε, μπορεί με, τα εθνικά κοινοβούλια όμως μπορούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε συνένεση όσον αφορά τις λύσεις και προσεγγίσεις που θα μας επιτρέψουν τη βελτίωση της εφαρμογής των συστάσεων αυτών. Κάποιες ομάδες το θέλουν αυτό. Πιστεύω ότι είναι θεμελιώδη σημασία σε αυτό το διάλογο που διεξάγεται με τα Εθνικά Κοινοβούλια να συζητήσουμε τρία ζητήματα. Μεταρρύθμιση της αγοράς εργασία γύρανση του πληθυσμού, δηλαδή το δημογραφικό θέμα, και οι επενδύσεις στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, γνωρίζουμε και το βλέπουμε ότι στα κράτη-μέλη γίνεται λόγος για την ψηφιοποίηση, για τις τεχνολογικές αλλαγές και μεταρρύθμισαν και μεταμορφώνουν ριζικά τις αγορές εργασίας αυτές οι αλλαγές. Διάφορες μορφές εργασίας διαφαίνονται και η αλλαγή εργασία γίνεται κάτι συνηθισμένο τώρα από ένα είδο εργασία ε, σε άλλη εργασία. Είναι μια πρόκληση, διότι η αγορά εργασία χρειάζεται ευελιξία από του ανθρώπου. Είναι πρόκληση για τα εθνικά κοινοβούλια και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να θεσπίζουμε νόμου που το καλύπτουν αυτό. Να απομακρυνθούμε από τα πτυχία, τα πανεπιστημιακά φερρυπίν και να, να επικεντρωθούμε επί των δεξιοτήτων. Πώ θα τι διαχωρίσουμε. Χρειάζεται επαγγελματική κατάρτιση, διαβίου, εκμάθηση, ε, Εξυγχρονισμό των γνώσεων και υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν εκτός αυτού του συστήματος. Θα πρέπει και αυτά τα άτομα να ενταχθούν και να μπορούν να περάσουν από τη μια δουλειά στην άλλη και να μπορούν να εργαστούν. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του δημόσιου τομέα, πρέπει να λάβουμε υπόψη εκεί τα χρήματα που χρειάζονται για την κάλυψη της γύρανσης του πληθυσμού. Υπάρχει αλλαγή δημογραφική και πιέζει τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μας. Αφορά όλα τα κατημέλη. Γύρανση τι σημαίνει, ότι αυξάνονται οι συνταξιούχοι. Και απ' την άλλη μειώνεται ο ενεργός πληθυσμός. Αυτό μακροπρόθεσμα δεν είναι κάτι βιώσιμο. Δεύτερη προτεραιότητα των κρατών μελών και όλων μας είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Πάνω απ' όλα εκεί που υπάρχουν πολλά χρέη, τεράστιο δημόσιο χρέος, όπως στη χώρα μου και στο, στο Βέλγιο και αλλού όπου υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες οι συντάξεις δεν μπορούν να καλυφθούν, η χρηματοδότηση των συντάξεων. Και αυτό είναι σημαντικό, έχει αντίκτυπο. Έχει αντίκτυπο στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, χρειαζόμαστε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις όσον αφορά την, την αγορά των κεφαλαίων και πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις δημόσιες επενδύσεις. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις επενδύσεις στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε μεγάλη ε, χαρά τις παρατηρήσεις. Κοιτάξτε, δεν, δώσατε, ξεκινήσαμε το καλό παράδειγμα, να δούμε τι θα γίνει με τους εθνικούς κοινοβουλευτές. Ε, Αλμπέρτο Ριμπόλα και Γιάζεκ σε ετοιμάζεται μετά. Ο κύριος Αλμπέρτο Ριμπόλα για την Ιταλία από τη Λέγκα του Βόρα έχει το λόγο. Το μικρόφωνο του δυστυχώ δεν ε, συνεδριάζουμε εδώ για να συζητήσουμε τα θέματα των οικονομικών πολιτικών στην Ευρώπη, ενώ στη Ρώμη αυτέ τι ώρε ξεκινάει η συζήτηση όσον αφορά ε, το θέμα του υπολογισμού και το, το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικού που τελεί βάση για τον επόμενο προπολογισμό, ε, που θα είναι η πρώτη κίνηση του, ε, τη νέα κυβερνήσεω. Και σκέφτομαι τι γίνεται σε διάφορε έδρε, πώ θα αντιδράσουν στη νέα στρατηγική για μεταρρυθμίσει που θα παρουσιάσει η Ιταλική κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Αντιπροέδρου Βάλτη Ντομπρόφσκη και, του κυρίου Μοσκοβιτσί, του, του Επιτρόπου Οικονομικών πιστεύουν ότι οι στόχοι ε, που έχουμε καθορίσει για τον ε, ε, κατά πρώτον φαίνεται ότι παραβιάζουν την, την πορεία προσαρμογής στην Ιταλία που έχει καθοριστεί. Ζήτησαν από την Ιταλική κυβέρνηση οι επίτροποι να εξασφαλίσουν ότι το νομοσχέδιο του προπολογισμού που θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα πρέπει να συνάδει με τους κοινού δημοσιονομικούς κανόνες. Στην Ιταλία όμως ξέρουμε ότι έχουμε ε, μπει στο Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη 22 Νοεμβρίου που πέρασε πριν από την σχηματισμό τη κυβερνήσεω αυτή, η Ευρωπαϊκή Περιτροπή θέτησε για μα την έκθεση όσον αφορά το μηχανισμό του κατάλληλου. Αν θέλετε διερμηνεί να σα μεταφράζουν αυτό λεξί, θα πρέπει να μιλάτε λίγο πιο αργά, λέει η κυρία Πρόεδρο. Καλώ. Αν μου δώσετε περισσότερο χρόνο, 30 δευτερόλεπτα περισσότερα. καλός. Πάνω απ' όλα θέλω να υπογραμμίσω ότι εκπροσωπώ μια κυβέρνηση που είναι υπεύθυνη, που θέλει να σέβεται τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στην Ευρώπη. Εκπροσωπώ και μια κυβέρνηση όμως γενναία, θαραλέα, που θέλει να θέσει ξανά στο επίκεντρο της Ευρώπης τους λαούς και τις απαιτήσει των λαών. Όχι μόνο τους αριθμούς και τη λιτότητα. Τα μέτρα, τα περιοριστικά που μας ενδιέφεραν κατά τη διάρκεια της εποχής της κρίσης, κατά την εποχή του Μόντι, την κυβέρνηση Μόντι, οδήγησαν σε ανεργία, φτώχεια και κοινωνική ανέχεια. Και δεχτήκαμε τα αποτελέσματα της ύφεσης πλήρη, χωρίς να μειώσουμε το δημόσιο χρέος όπως θέλαμε. Αντίθετα, συνεχώς αναπτύχθηκε και ξεπέρασε το 130% του ΕΠ. Υπό το φω τέτοιων αποτελεσμάτων, αυτή η πολιτική αποκλειστική λιτότητα θα πρέπει τώρα να αποθηκευτεί, να, να, μπει, να την αφήσουμε εκτό. Διαβάζω με χαρά το σχέδιο ψηφίσματο, όπου απευθύνει έκκληση για περισσότερη ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη, ούτω ώστε να επαναπροωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ίδια η ανάπτυξη. Ε, για αυτό το σκοπό ζητούμε να επικαιροποιηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, όχι μόνο για το κομμάτι που αφορά τη σταθερότητα των δημοσιονομικών, αλλά και για το θεμελιώδες θέμα της ε, ανάπτυξης. Ε, η Ιταλία σήμερα παραμένει ε, στην τελευταία σειρά της ανάπτυξης από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, άρα είναι σωστό η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου που σήμερα εκπροσωπώ να υποστηρίξει τη νέα οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Πρόκειται περί φιλόδοξου προγράμματο οικονομική πολιτική που έχει σαν στόχο πάνω απ' όλα να ανταποκριθεί στην αύξηση τη στόχια που καταγράφηκε από την κρίση και μετά, κυρίω μεταξύ των νέων και πολυμελών οικογενειών, και να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τι συντάξει, δημιουργώντα περισσότερο περιθώριο για την απασχόληση των νέων, εγγυόμενη έτσι την πλήρη βιωσιμότητα οικονομική των συστημάτων προνοία. Αυτοί οι στόχοι πρέπει να συνδυάζονται με αυτόν που η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι η απόλυτη προτεραιότητα για τη χώρα, δηλαδή την επαναπρόθεση τη βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύσει, απασχόληση και τη μείωση των ανισοτήτων και ζήτησε εξάλλου στο σχέδιο ψηφίσματος του Κοινοβούλου. Ε, ο ελιγμό αυτό τη Ιταλία θα, θα τονώσει την οικονομική δραστηριότητα που θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εκτιμήσετε δημοσιονομικά δεν συμπεριλαμβάνονται αναδραστικά τη μεγαλύτερη ε, αύξηση στον προπολογισμό. Το μεγάλο υψηλότερο επίπεδο του ΑΕΠ του ονομαστικού θα μειώσει τη σχέση χρέου ΑΕΠ κατά τη διάρκεια τη Τριετία. Και κλείνω. Αυτό το πρόγραμμα μεταρρύθμιση πέραν αυτού καλύπτει όλε τους ε, του τομεί των τεσσάρων συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όμω χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο εύρο και διαφοροποιείται σε κάποια σημεία επί τη ουσία όσον αφορά τι προτεραιότητε από τη μείωση του φορολογικού βάρου, όπω επηρεάζει την εργασία, μέχρι την ανάδυση τη ε, υποβόσκουσα οικονομία και να καταργηθούν οι αδικίε και η διαφθορά. Νέα μέτρα στον τραπεζικό τομέα, αν θέλετε να ολοκληρώσετε, διότι ξεπεράσατε ήδη το χρόνο σα, λέει Πρόεδρο. Κανονικά είναι τρία λεπτά. Ήδη είσαστε τέσσερα λεπτά, αν έχετε την καλοσύνη. Καλώ, δάτομαι με τη ευκαιρία για να υπογραμμίσω στα πλαίσια τη συζητήσεω του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου τη σημασία να έχουμε ποσοστό σημαντικό των πόρων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στι πολιτικέ που τονώνουν την ανάπτυξη που θα συνοδεύουν τι εθνικέ πολιτικέ. Διαβάζω με, με, με ικανοποίηση ότι δεν θα περικοπεί η πολιτική συνοχή, που είναι σημαντική πτυχή για τι επενδύσει. Και πιστεύω ότι δίπλα από τα ποσά για τι νέε πολιτικέ θα πρέπει να δεθεί μεγαλύτερη προσπάθεια, καταρχήν μεγαλύτερη προσπάθεια για να εγγυηθούμε ήδη τη χρηματοδότηση που προβλέπεται για πιο παραδοσιακέ πολιτικέ, ξεκινώντα από την κοινή αγροτική πολιτική. Αγαπητέ συνάδελφε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, μη διαβάζετε πολύ γρήγορα και δεύτερον, τηρήστε το χρόνο μιλία σα και θα έχουμε τέτοια απόκληση που στο τέλο οι τελευταίοι δεν θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο. Ε, θα, θα γίνω πιο αυστηρή για τα τρία λεπτά και κάτι, αλλά και κάτι. Λοιπόν, Πολωνία, ο κύριος Γιάζικ Βοσόφσκι του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνης και κατόπιν ο Μιγγέλ Γκίγκας εκ μέρους της ΓΚΟΕ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, κύριε Βοσόφσκι, έχετε τον λόγο. Κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να μην διαβάζω την ομιλία μου. Στην Πολωνία λέμε ότι καλύτερα να μιλάει κανείς ε, από, το, στήθους. Δύο λόγια σχετικά με την επερχόμενη εφταετή περίοδο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο μελλοντικό προπολογισμό της ε, η Πολωνία θα ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις μας, αλλά θα μας δώσει και πόρους για την, ικανοποίηση, για την κάλυψη των μελλοντικών ε, δεσμεύσεών μας. Σημαντική για μας είναι η ΚΑΠ. Το μείον 10% που προτάθηκε, ενδεχομένω δεν είναι η καλύτερη λύση. Μείωση της συνοχής κατά 46%. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Για μας η πολιτική συνοχή ένα στόχο έχει. Ο στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν μικρότερες δυσαναλογίες και ανισορροπίε ανάμεσα στι διάφορε οικονομίε. Θέλουμε δηλαδή να τηρηθούν τα κριτήρια σύγκληση. Αν προχωρήσουμε έτσι θα πετύχουμε. Τώρα, οι νέε προκλήσει. Οι νέε προκλήσει δυστυχώ κάποιε από αυτέ οφείλονται σε κάποιες ατυχείς πολιτικές αποφάσεις κάποιων κρατών μελών. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Αναφέρομαι στη μετανάστευση, στην εσωτερική ασφάλεια και την εξωτερική ασφάλεια. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε πόρους για την προστασία αυτών των τομέων. Προτείνουμε την το νέο πρόγραμμα, το Invest EU, που ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Θεωρώ ότι για οποιαδήποτε επιχείρηση, σε οποιαδήποτε χώρα θα αποτελέσει μια τεράστια ευκαιρία. Ε, πώς έχουν τα πράγματα. Ανάπτυξη κατά 1,11% ή μάλλον το 1,11% είναι το επίπεδο που ε, ε, αυξάνει ελάχιστα σε σχέση με τα τωρινά. Δεν το θεωρούμε παρκές. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ υπερβολικά παθητική προσέγγιση. Δεν είναι αρκετά ε, φιλόδοξη και η Πολωνία είναι διατεθειμένη να το αλλάξει αυτό. Έτσι θα θέλαμε να ξεπεράσουμε το 1,11% του αέπα θα θέλαμε να προσεγγίσουμε περισσότερο το 1,2%. Υπό την άποψη αυτή θα μπορούσαμε τελικά να χρηματοδοτήσουμε τις περισσότερες προκλήσεις, τις υφιστάμενες αλλά και τις μελλοντικές. Είναι λοιπόν αρκετά προφανές ότι η προσέγγιση της χώρας μου διαφέρει από τις προσεγγίσεις των άλλων χωρών. Θέλουμε να προχωρήσουμε και να αυξήσουμε, όχι να μειώσουμε την εθνική συμμετοχή. Θεωρούμε ότι για να εκμεταλλευτούμε όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να κινούμαστε προς την ε, ε, κατεύθυνση αυτή αλλά οι πόροι που έχουν συγκεντρωθεί να, ε, να χρησιμοποιούνται ορθολογικά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ο Μιγέλ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ΓΚΟΕ. Ε, θα μιλήσω πορτογαλικά, λέει ο μιλητής. Και θα είμαι σύντομος, θα μιλήσω σε, ε, μόνο για τρία λεπτά. Θέλω να εκφράσω τις ανησυχίες μας για το ευρώ και την πολιτική, τις πολιτικές της Ευρωζώνης. Βεβαίως έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα της Ευρωζώνης, δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, Μοιάζει ότι το ευρώ προκαλεί ε, εκφύσεως λιτότητα. Δεν επιτρέπει την λειτουργία των εθνικών σταθεροποιητών, των φυσικών σταθεροποιητών και διάφορες χώρες ε, ε, αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν πολιτικές που ενισχύουν τον οικονομικό κύκλο. Το ισχυρό ευρώ δεν είναι καλό για τις οικονομίες της περιφέρειας της ε, Ευρωζώνης. Κυρίως για τα μη εμπορεύσιμα αγαθά, δηλαδή τα ακίνητα και ο τουρισμός που μοιάζει ότι είναι οι δύο μόνοι τομείς που αναπτύσσονται και οδηγούν σε ανισορροπίες. Και αυτά δεν έχουν επιληθεί από την Ευρωζώνη. Τα, ε, οι λύσεις έρχονται μέσω ε, του γεγονότος ότι οι εργαζόμενοι στις περιφερειακές οικονομίες δίνουν το αίμα τους. Παρά τα αυτά, το μόνο που άλλαξε από την κρίση είναι ότι τώρα μοιάζει ότι βρισκόμαστε στην άνοδο του οικονομικού κύκλου. Μοιάζει ότι υπάρχει αύξηση των επιτοκίων, αυξάνονται οι τιμές του, του πετρελαίου. Είναι σαφές ότι τώρα ε, εμφανίζεται μια νέα κρίση οι οικονομίες λοιπόν της περιφέρειας πρέπει να αποφύγουν την, να παγιδευτούν στην λεγόμενη ευρώ παγίδα. Το πρόβλημα μοιάζει ότι είναι ότι η οικονομία εξυπηρετεί το ευρώ και όχι το ευρώ την πραγματική οικονομία. Ένα βασικό θέμα στην Πορτογαλία είναι η ανάκαμψη της ε, νομισματικής κυριαρχίας. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλουμε να ξαναρχίσει η ανάπτυξη της οικονομίας και στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες περιφέρειες που έχουν υποφέρει στο διάστημα αυτό. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Μαργαρίτα Μάρκες από την Πορτογαλία. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ορίστε. Και πάλι η Πορτογάλος ομιλητής από το Εθνικό Κοινοβούλιο αυτή τη φορά. Θα ήθελα να θέσω κάποια θέματα, αν μου επιτρέπει ο χρόνος. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος ε, έκανε μια καλή σύνοψη της έκθεσης που μόλις ε, διαβάσαμε. Φυσικά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι σημαντικό εργαλείο για την εσωτερική πολιτική της Ένωσης έχουμε παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυ τις εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και νομίζω ότι σήμερα αντιμετωπίσουμε σοβαρή πρόκληση, η οποία συνίσταται στην εξέβριση της σωστής ισορροπίας ανάμεσα σε δημοσιονομικές πολιτικές που να είναι υγιείς και στις ε, επενδύσεις και από την άλλη την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Η ισορροπία θα στηριχθεί σε, μια, σε έναν όρο. Ευελιξία. Ευελιξία κατά τη δική μας έννοια όμως, που είναι το αντίθετο από το να είναι κανείς χαλαρός. Η ευελιξία πρέπει να καθοριστεί ξεκάθαρα στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Δεν θα πρέπει να είναι κάτι που ερμηνεύεται απλώς κατά το δοκούν από του εκπροσώπου των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Θα αναφερθώ στην περίπτωση Πορτογαλία, η οποία αποτελεί ένα παράδειγμα, θα έλεγα, καλό παράδειγμα. Μια αναπτυσσόμενη οικονομία που άφησε τη χώρα, επέτρεψε στη χώρα να τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της ε, Ευρωζώνης. Είδαμε μείωση των ανισοτήτων και αύξηση των επενδύσεων, έστω και με τρόπο αρκετά εύθραυστο έχουμε ανάκαμψη. Αν δούμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το ευρωπαϊκό εξάμεινο, το θέμα που τίθεται είναι πώς μπορεί ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών ε, Δικαιωμάτων να ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ο πυλώνας των, ευρωπαϊκών, ε, των κοινωνικών δικαιωμάτων θα ενισχυθεί μόνο αν ενσωματωθεί σωστά στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τρίτον, πρέπει να ενστερνιστούν τα κράτη-μέλη τις συστάσεις αναχώρα. Μιλάμε για κοινή κυριαρχία. Το θέμα του να ενστάνεται κανείς ε, ιδιοκτησία, να ενστερνίζεται τις συστάσεις αυτές, είναι ακριβώς αυτό ε, το θέμα αν δούμε την υλοποίηση των κανόνων, αυτοί εφαρμόζονται από τα εθνικά θεσμικά όργανα και θα πρέπει λοιπόν τα εθνικά κοινοβούλια να καταβάλουν προσπάθεια να συνεργαστούν με τις πολιτικές δυνάμεις, τα πολιτικά κόμματα, ε, στις κυβερνήσεις που είναι κυβερνήσεις ε, που υποστηρίζονται από περισσότερα από ένα κόμματα, κυβερνήσεις συνασπισμού. Χρειαζόμαστε περισσότερη κοινοβουλευτική δημοκρατία σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, λέει στα πορτογαλικά ο πρόεδρος. Ουντέ Καλούνε. από την Εστονία, ομάδα της των φιλελευθέρων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, θα μιλήσω Ιταλιστή. Ξεκινώντας θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου, διότι εδώ υπάρχουν τέσσερις χώρες που είναι λιγότερο ίσες απαλές, που δεν, έχουν, δεν μπορούν να μιλήσουν στη γλώσσα τους. Ελπίζω είναι η τελευταία φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Τώρα στρεφόμενοι προς το επιχείρημα το σημερινό, το θέμα το σημερινό, την οικονομία, με ανησυχεί διότι δεν μιλάμε για τη μεταρρύθμιση την πιο σημαντική, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση του Μάστικ βασίζεται στην αρχή της συγκράτησης του πληθωρισμού που επικρατεί έναντι ουδήποτε άλλου στοιχείο και όχι επιπλήρου απασχόληση. Όσο παραμένει αυτή η αρχή, οι οδηγίε που στα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση των ισοτήτων κλπ. κλπ ε, ε, δεν μπορούν να επιτευχθούν. Ο πληθωρισμό πάντα είναι φίλο ε, του, του εκείνου που χρωστάει και όχι εκείνου που, που πιστώνει. Είναι εχθρό των εισαγωγείων και φίλο των εξαγωγείων εάν δεν υπάρχει για άλλους εργασία, το γεγονός ότι ο άνεργος πρέπει να βρει μια σημαίνει ότι θα πρέπει να χάσει θέση του αυτός που έχει τη θέση απασχόληση με αυτόν τον τρόπο. Ο μηχανισμός είναι αυτός που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να επιβάλλει. Και έτσι έχουμε μια αντικατάσταση ενός ε, εργαζομένου ε, από έναν άνεργο και πέφτει η αμοιβή. Και έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι φίλη της συμπίεσης των μισθών. Και αυτή θα πρέπει να αλλάξει σαν πολιτική. Θα πρέπει να, να δώσουμε χώρο στα κράτη-μέλη, περιθώριο στα κράτη-μέλη, για να βοηθήσουν τις επενδύσεις, ούτω ώστε να είναι στοχευμένες επενδύσεις. Εν, εν πρώτης, οι επενδύσεις να αφορούν την πλήρη απασχόληση. Χρειάζεται σχεδιασμός των επενδύσεων, που θα έχουν στόχο ε, εκεί που μπορεί να επιτευχθεί ε, η σωστή οικονομική απόδοση. Χρειάζεται εργασία για όλους. Μόνο έτσι θα φτάσουμε στην ανάπτυξη, ευημερία και ισότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για τα έξοχα Ιταλικά σας. Δεν μπορώ να ζητήσω συγγνώμη. Δεν φταίμε εμείς που δεν έχουμε όλες τις γλώσσες διαθέσιμες σήμερα. Είναι τεχνικά θέματα που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και υποστηρίζουμε την πολυγλωσία ένθερμα. Και πάντα στενοχωρούμεθα πολύ όταν δεν μπορούμε να παράσχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Ευτυχώς όμως ήσασταν πολύ ικανοί να κάνετε αυτή την ομιλία που ήταν πιο ευπρόσδεκτη για τους σοσιαλιστές από ότι για τους φιλελεύθερους. Αυτές είναι έννοιες που δεν ακούμε πάντα τους φιλελεύθερους φίλους μας, συναδέλφους μας. Ευτυχώς επίσης η επικράτηση της σταθερότητας των τιμών έναντι της οικονομικής αναπτύξεως δεν είναι επικράτηση. Είναι ο πρώτος το στόχος της νομισματικής πολιτικής, όχι της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης. Αληθεύει αυτό που είπατε, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, ασχολείται με την νομισματική πολιτική, τη σταθερότητα της τιμής είναι πρώτη το στόχος. Και η ΕΚΤ έδειξε όμως ότι μπορεί να πετύχει άλλους στόχους. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, Στη συνθήκη δεν λέγεται ότι η σταθερότητα των τιμών επικρατεί είναι ισχυρότερη από την ανάπτυξη. Εμείς που διαμορφώνουμε την πολιτική προσπαθούμε να συμφιλιώσουμε τους δύο αυτούς ε, στόχους. Και αυτό συζητούμε σήμερα. Επόμενος, για το Ευρωκοινοβούλιο. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης. Έχετε το λόγο. Απουσιάζει. Θα μιλήσει αργότερα όταν επιστρέψει ο κ. Παπαδημούλης. Ο κ. Μπαλούρα από την Ελλάδα, Γκουε, NGL, Ενωτική Αριστερά, καλώ ήρθατε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Έχετε δώσει αγώνες για την χώρα μου, την Ελλάδα και θυμίζω ότι για πρώτη φορά συμμετέχουμε σαν ισότιμοι συνομιλητές ε, στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μέχρι τώρα, επειδή είμαστε τα μνημόνια, ε, είμαστε απλώς παρατηρητές. Περάσαμε δηλαδή 8 χρόνια με βάσανα, πόνο και μεγάλη ανεργία, καταβήθηση του ΑΕΠ. 25% του εθνικού μας πλούτου χάθηκε σε αυτά τα μνημόνια, τα οποία γίνανε με λαθεμένες πολιτικές και λαθεμένες συνταγές. Ε, τώρα πάει η οικονομία καλά, τα βάσανα όμως και πληγές παραμένουν. Το πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκή και Νοσματική ε, Ένωση, συνάδελφοι, χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλειοθήκη της νεοφιλελεύθερης ατζέντα. Ιδιωτικοποίησης, καταστροφή του κράτους πρόνοια, τα υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής από τις οικονομικές ελίτ και η κατάρριση των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων οδήγησαν σε μεγαλύτερη απόκληση μεταξύ των κρατών μελών και περιφερειών και μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες πλήττοντας την εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή. Έχω την εντύπωση κύριε Πρόεδρε ότι είναι σαν να βρισκόμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο, στο, στο Τιτανικό και άλλοι άδουν, τραγουδούν, άλλοι χορεύουν και άλλοι είναι στα μπάρια, αλλά όλοι μαζί θα βυθιστούν. Εάν δεν προσέξουμε, πού πάμε. Για παράδειγμα, θέλουμε ένα σύμφωνο απασχόληση, όπως είπατε σωστά προηγουμένως, απαντώντας στην συνάδελφό μας από την Εστονία, για την απασχόληση στην ανάπτυξη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο επίση υπενηχθήκατε, να έχει και άλλους στόχους και όχι μόνο την προστασία από την ανάνοδο των τιμών. Θα πρέπει να υπάρχουν συλλογικέ διαπραγματεύσει και συλλογικέ συμβάσει εργασία. Θα πρέπει να σεβόμαστε το δικαίωμα στην απεργία. Θα πρέπει να υπάρξει αναθεωρημένος ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης που θα ενισχύει την κοινωνική και οικονομική σύγκληση και συνοχή μεταξύ των λαών για να καταπολεμηθεί και το κοινωνικό ντάμπινγκ. Θα πρέπει να, ε, να υπάρχει σχέδιο κοινωνικών επενδύσεων μια ολοκληρωμένη στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής προστασίας. Θα, θα υπάρξει ρήξη με τις πολιτικές συλλητότητες που είναι επιζήμιοι για τους αλλούς λαούς της Ευρώπης και συμβάλλουν στην ξενοφοβία και στην άδοδο των ακροδεξιών δυνάμεων. Και τέλος θέλω να πω κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει αυτά τα κράτη τα οποία ε, μπήκανε σε καθεστώτα έκτατης ανάγκη να τα θεωρήσουμε ως τέτοια και να ε, δώσουμε δυνατότητες ενός πλαισίου που θα δημιουργηθεί για την υποστήριξη της οικονομίας, αυτό δηλαδή που έχουν μπει στα μνημόνια και είναι 4-5 κράτη. Τέλος, μια διεθνή σύνοδος κορυφής στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό τον καθορισμό ενός οδικού χάρτη και ενός κοινού σχεδίου δράσης για τον τερματισμό των φορολογικών παραδείσων και της φοροδιαφυγής ε, ο, ο, ο εισηγητής, ο κύριος Μαυρίδης, είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Αναφέρω ένα, την εγγύηση καταθέσεων. Και η χώρα του έχει πληγεί από αυτήν την ιστορία και πιθανόν να πληγούν και άλλα κράτη. Και τέλο, αύξηση του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίο θα επικεντρωθεί ειδικά στην κοινωνική ανάπτυξη και στην ανωδική κοινωνική σύγκληση, εισάγοντα και πάλι την έννοια τη πολιτική συνοχή ανταποκρινόμενη στι ανάγκε του κάθε κράτου μέλου. Κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδυσία, διαφάνεια και εποπτεία των ευρωπαϊκών πολιτικών και θεσμών, ενδυναμώνοντας το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Grazie. Um, Ευχαριστώ πολύ θα ήταν ενδιαφέρον, αλλά ίσω ο κ. Παπαδημούλης ε, θα μπορούσε να μα πει λίγο περισσότερα για αυτήν την ε, θετική για μένα, αλλά γενικότερα για τη στρατηγική, για το πώ ενδεχομένως να μην εφαρμόσετε κάποια μέτρα που είχαν ζητηθεί αρχικά στον προπολογισμό σας. Ενδιαφέρον θέμα για να συζητήσουμε ε, στο, πλαίσιο αυτό, αλλά αν έχουμε το χρόνο. Επόμενος ομιλητή, ο κύριος Νεοφίτου από το Κυπριακό Κοινοβούλιο, ε, ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Παρακαλώ. Και η χώρα μου πέρασε από μνημόνια. Δεν αντικρίσαμε τις συστάσεις αλλά και το μνημόνιο ως τιμωρία, αλλά ως μια ευκαιρία να διορθώσουμε τα του οίκου μας και να αντιμετωπίσουμε τη δημοσιονομική και την τραπεζική κρίση. Σήμερα η χώρα μου είναι εκτός μνημονία και από τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα η οικονομία βρίσκεται σε ένα θετικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης από τους ψηλότερους της Ευρώπης με δημοσιονομικά πλεονάσματα που ξεπερνούν το 3%. Μια ανεργία που έφτασε το 2013 στο 18% είναι σήμερα κάτω από το 7, γύρω στο 7% και ευελπιστούμε ότι σε δυο περίπου χρόνια η κυπριακή οικονομία θα είναι μια οικονομία με πλήρη απασχόληση. Παράλληλα παρατηρούμε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2018 και αυτές δεν τις αντιμετωπίζουμε ως κάτι που κάποιος θα θεωρούσε ως τιμωρία αλλά θέλουμε αυτές τις συστάσεις να τις υλοποιήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και το συντομότερο δυνατόν. Ήδη η τρίτα σύσταση που αφορούσε την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσα από κινήσεις του τραπεζικού συστήματος τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες έχουν μειωθεί δραστικά όπως επίσης και η αλλαγή που είναι η δεύτερη σύσταση του πλαισίου αφαιρεγγιότητος έχει βελτιωθεί τον περασμένο Ιούλιο. Χρειάζονται όμως οι μεταρρυθμίσεις όπως η σύσταση η πρώτη για πιο αποτελεσματική δημόσια υπηρεσία και παραγωγικό δημόσιο τομέα, η τέταρτη σύσταση για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση αλλά και βελτίωση των επιδόσεων των κρατικών εταιριών. Αλλά δεν είμαι αισιόδοξο αν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αποκρατικοποιήσεις. Σημειώνουμε επίσης τη σωστή επισήμανση και σύσταση της Επιτροπής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ανέργων νέων μας και όσον αφορά την έκτη σύσταση για την υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας μέχρι το 2020 είμαστε πεπισμένοι και σίγουροι ότι αυτό θα το κατορθώσουμε αφού το πρώτο στάδιο θα εφαρμοστεί από την 1η Μαΐου του 2019. Η Κύπρος ξεπέρασε την κρίση, την αντιμετωπίσαμε ως μια ευκαιρία, μια μεγάλη πρόκληση να γίνουμε καλύτεροι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενο ομιλητή από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Περβάνος Μπερέζ, ε, Σοσιαλιστική Ομάδα. Ευχαριστώ αυτή η ανταλλαγή μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη φάση του οικονομικού κύκλου είναι πάντα ενδιαφέρουσα. Γιατί όπως είπα όταν προέδρευα, τώρα που τα εθνικά κοινοβούλια προσπαθούν να εγκρίνουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς και που εμείς θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα βασικά θέματα του επόμενου οικονομικού κύκλου, είναι κατάλληλο να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Υπάρχουν δύο-τρία θέματα που νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν όλους. Όπου αν λοιπόν υπάρξει μια συμμαχία μεταξύ Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Το πρώτο θέμα είναι πώς αξιοποιεί και αν αξιοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα εργαλείο πολύ πολύτιμο, το οποίο και εμείς συμβάλαμε να υπάρξει, τη διαδικασία μακροοικονομικής ανισορροπίας δεν τολμάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει αυτή τη διαδικασία πλήρω οπότε δεν έχει και κανένα αποτέλεσμα. Και αυτό σημαίνει ότι διατηρούνται οι ανισορροπίε μεταξύ των χωρών που έχουν πλεονάσματα και των χωρών που έχουν ελλείμματα και δεν διορθώνεται αυτή η κατάσταση. Και τι διαπιστώνουμε. Πέρα από τις ε, εντάσεις ε, μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης θα μπορούσε τελικά να καταλήξει και σε εντάσεις μεταξύ της Ευρωζώνης και των υπολείπων χωρών και του υπολείπου κόσμου. Δεν είμαι φυσικά ο του Ντόναλτ Τραμπ. Αλλά όταν ο Ντόναλτ Τραμπ λέει ότι κάποιες ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν πολλές εξαγωγές γιατί με αθέμητο τρόπο εποφελούνται από αυτά τα πλεονάσματα που δεν διορθώνονται εντό της Ένωσης όπου παράγονται αυτό είναι σοβαρό θέμα. Δεν βλέπω πόσο χρόνο έχω. Έχω χρόνο λοιπόν να αναφερθώ και σε ένα δεύτερο σημείο. Ε, καλά, να υπερβώ λίγο το χρόνο μου. Να ασχοληθώ με ένα άλλο θέμα που θεωρώ ιδιαίτερος ουσιώδες. Είναι τα προγράμματα που εκπονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου ορισμένα θέματα που μας απασχολούν μόνιμα μπορεί να επανέλθουν στο προσκήνιο είναι η συζήτηση για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Πρόκειται για παγίδα που θα πρέπει να αποφευχθεί. Τώρα το θέμα δεν είναι να καταδικάζουμε και να επενούμε, να λέμε ο ένας τα πάει καλά, ο άλλος είναι σκάρτος. Πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον κοινό μας πλούτο, που είναι το ευρώ. Και αυτό είναι το τρίτο θέμα που θέλω να αναφέρω. Βλέπουμε ότι σε ορισμένες χώρες, αλλά και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ορισμένες φορές υποκύπτουμε στον πειρασμό να θεωρήσουμε το ευρώ υπεύθυνο για όλα τα προβλήματα και όλες τις καθυστερήσεις των οικονομιών μας. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι παντού όπου οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να βγουν από το ευρώ, βλέπουμε ότι υπάρχει αντίδραση, αντίσταση, γιατί θα ήταν τρομερό το κόστος και δεν υπάρχει κανένα πολιτικό πρόγραμμα που να μπορέσει να υποσχεθεί ένα ε, ευτυχές μέλλον για το λαό παράλληλα επιδιώκοντας την έξοδο από τον Ευρωπαϊκό. Πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι για να δούμε ποιου κανόνες πρέπει όλοι να τηρούμε για να μπορέσουμε να αποφεληθούμε όλοι από αυτό το νόμισμα. Και αυτό πρέπει να, να επιχειρήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο εγγυσμένο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο και τώρα, ο κύριος Σκόπετσεκ από την Τσεχία και την ομάδα ECR. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, από ό,τι άκουσα από τους προηγούμενους ομιλητές, μου δημιουργείται εντύπωση ότι σχεδόν κανείς δεν ε, έχει αντιληφθεί ότι στην Ευρώπη ζούμε υπεράνω των δυνατοτήτων μας. Άμα δούμε πόσες χώρες έχουν μόνιμα ελλείμματα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση να ξοδέψουμε και τις τελευταίες οικονομίες μας στην ουσία. Στα κείμενά σα λέτε ότι πρέπει να είναι στοχευμένη η δημοσιονομική μας πολιτική. Τι σημαίνει αυτό. Θέλουμε οι προπολογισμοί μα να δημιουργήσουν περαιτέρω ελλείμματα γιατί αυτός είναι ο λόγος που δημιούργησε και ενέτεινε την ε, κρίση και στην Ευρωζώνη και ευρύτερα στην Ευρώπη από το 2008. Ο Τιτανικός που λέγεται Ευρώπη, όπως ανέφερε και ένας προηγούμενος ομιλητής, δεν προέκυψε επειδή είχαμε σωστά προγραμματισμένους προπολογισμού προέκυψε επειδή είχαμε κράτη προνοίας τα οποία δεν ήταν χρηματοδοτήσιμα. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες τώρα να χαλαρώσουμε κάποιους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και ακόμη και κάποιες ιδρυτικές χώρες της Ευρωζώνης δεν σέβονται τους κανόνες που οι ίδιες θέσπισαν. Και δεν σέβονται τους κανόνες που οι ίδιες αυτές χώρες απαιτούν άλλες χώρες να σέβονται. Χώρες που ε, επιδιώκουν να μπουν στην Ευρωζώνη, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ιδιωτικό τομέα παράγει πλούτο. Εάν δημιουργούμε όλο και περισσότερου κανονισμού, δεν θα δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία στην Ισπανία, στην Ιταλία, σε όλε τι άλλε χώρε, όπου υπάρχει τεράστια ανεργία, κυρίω των νέων. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να θέτει, να είναι παράδειγμα για τον κόσμο. Τώρα που συζητάμε το επόμενο πολιτέ διομισονικό πλαίσιο και στην Τσεχία, συζητάμε το θέμα αυτό στο κοινοβούλιο μα και καλούμε την Ένωση να κάνει οικονομίε. Γιατί όταν θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να μειωθεί, όχι να αυξηθεί ο προπολογισμό. Δεν θα πρέπει να αυξήσει η Ένωση του ίδιου πόρου τη. Θα πρέπει να κάνει εξοικονομήσει. Γενικά είμαι ιδιαίτερα επικριτικός έναντι ε, κάθε απόπειρα να, να εναρμονιστεί η φορολογία. Γιατί για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αυτό θα σήμαινε τέλος στην ανταγωνιστικότητά τους. Δεν έχουμε τόσο ευρείες αγορές όπως οι ε, παλιές χώρες για να αντιμετωπίσουμε ε, τον ανταγωνισμό για παράδειγμα της Γαλλίας θα ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για τις οικονομίες μας κάτι τέτοιο. Και τώρα, κάτι άλλο. Από όλες τις ε, πλευρές του πολιτικού φάσματος, από τους ελεύθερους μέχρι τους κομμουνιστές, ακούμε να λέγεται ότι το μόνο που θα πρέπει να γίνει η Ευρωζώνη το θα πρέπει να κάνει η Ευρωζώνη είναι ο καθένας να επιλέξει το επίπεδο ένταξής του στην Ευρωζώνη. Δεν είναι δυνατόν με τόσο ευρύ φάσμα απόψεων να φτάσουμε σε ένα συμβασμό. Τα κράτη-μέλη να επιλέγουν τι θα πρέπει να κάνει η κάθε χώρα. Εάν οι φίλοι μας οι κομμουνιστές θέλουν να πάνε κάπου αριστερά, ας το κάνουν. Εγώ από μια χώρα όπου έχουμε ε, βαθιά πείρα από κομμουνισμού και δεν θέλω να επαναληφθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζετε φυσικά ότι ε, από πλευρά της χώρας σας ακούμε και αυτούς που λένε ότι θέλουμε περιορισμένο προϋπολογισμό, δεν θέλουμε περικοπές ε, στις, στην πολιτική συνοχής και αυτά δύσκολα συνδυάζονται. Ε, αν έχει κανείς μικρότερο προπολογισμό ευρωπαϊκό, μπορεί, πώς μπορεί να μην έχει λιγότερα χρήματα για την πολιτική συνοχής. Ε, θα υπήρχε κάποια συνεκτικότητα στις, σε αυτά που λέτε. Αν Λοιπόν, η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Σίτο από τη Γερουσία της Ρουμανίας, εκπροσωπεί το ΕΛΚ. Θα μιλήσω, κύριε Πρόεδρε, για τις ε, αναχώρα συστάσεις, συστάσεις αναχώρα που ε, αφορούν τη Ρουμανία και τα θέματα που εφαρμόζει η κυβέρνηση της χώρας. Ξέρετε ότι το διαρθρωτικό έλλειμμα της Ρουμανίας θα αυξηθεί και οι συστάσεις σας θα γίνουν πιο δύσκολες να, δύσκολο να εφαρμοστούν. Το ερώτημά μου είναι γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν προσπαθούν να βρουν τρόπο να, προσπαθούν να κάνουν την κυβέρνηση να τηρήσει αυτές τις συστάσεις. Παρά το θέμα όμως αυτό που θέλω να θέσω είναι το θέμα του προβλήματος της, ε, του εργατικού δυναμικού στη Ρουμανία και στην Ανατολική Ευρώπη. Διότι με την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, που είναι σπουδαίο για τη Ρουμανία αλλά και για την Ευρώπη, αντιμετωπίζουμε τώρα ένα άλλο πρόβλημα στη χώρα μου. Προσπαθούμε να πετύχουμε την ανάπτυξη οικονομίας στο επόμενο διάστημα, αλλά έχουμε δυσκολία διότι περιορίζεται το εργατικό δυναμικό και δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους εργαζόμενους να επιστρέψουν σε εμά από την Ευρώπη ή άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Η μόνη λύση που μας απομένει λοιπόν είναι να εισάγουμε εργαζόμενους από χώρες εκτός Ένωσης. Όταν όμως το προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, διότι η εισαγωγή εργαζομένων από χώρες εκτός Ένωσης ε, ε, σημαίνει ότι αυτοί θα έχουν ε, διαφορετική μεταχείριση από ότι ε, οι εργαζόμενοι της χώρας, δηλαδή θα πληρώνονται περισσότερο. Προσπαθούμε λοιπόν να το ξεπεράσουμε αυτό το θέμα. Άρα, άρα πρέπει να επανεξετάσουμε αυτό το ρόλο κατά την, το κανόνα κατά την άποψή μας πρέπει να πληρώσουμε πάνω από το μέσο μισθό στους ε, εισαγόμενους εργαζόμενους, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να πληρώσουν τον μέσο μισθό. Η Ρουμανία και οι άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ε, θέλω να επισημάνω, αντιμετωπίζουν πρόβλημα εργατικού δυναμικού. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Ντεμπόνο από τη Μάλτα. Ε, προσωπεί την ομάδα ΕΛΚ. Sorry, my mistake. Έκανα λάθος, λέει ο πρόεδρος, με συγχωρείτε, η κυρία Ντεμπόνο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ την Επιτροπή που μας δίνει τη δυνατότητα ως εθνικούς βουλευτές να ανταλλάξουμε απόψεις ε, για το σχέδιο έκθεσης που αφορούν την CSR. Ε, Πιστεύω ότι ε, ε, θα είμαστε πολύ αποτελεσματικοί στη συζήτηση για, τις, ε, ε, για την ετήσια έκθεση και που τελικά επηρεάζουν τον προγραμματισμό του προπολογισμού κάθε χώρα. Γνωρίζω ότι η διαδικασία της αναδιάρθρωσης των κονδυλίων των, του Ταμείου Συνοχής είναι εν εξελίξει στην Επιτροπή. Τα ταμεία αυτά θα ενισχύσουν τις οικονομικές και κοινωνικές επενδύσεις. Η βιωσιμότητα και ε, παραμένει ένα θέμα στη χώρα μας παρά την εντυπωσιακή οικονομική μας ανάπτυξη. Παρά τα αυτά έχουμε ε, όλο και ε, ένα πληθυσμό που συνεχώς γερνά και έχουμε ψηλό επίπεδο πληθωρισμού και χαμηλή συμμετοχή γυναικών στο, στην εργασία. Παρά τα αυτά έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ανθρώπων που εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο. Ως εκ τούτου όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν μεγάλες δυσκολίες στην ε, στήριξη του των συστήματος συντάξεων. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι ένα ψηλό επίπεδο ζωής θα μπορεί να ε, ε, ισχύει για όλους εξίσου. Θέλουμε λοιπόν μια ολοκληρωμένη ισχυρή στρατηγική ώστε οι χώρες ε, όπως η Μάλτα που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έχουν μακροπρόθεσμα πρόβλημα στο συνταξιωτικό του σύστημα. Αυτό φυσικά θα είναι ε, ε, ένα θέμα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Παραμένουμε στη Μάλτα. Ο κύριος Bedingfield έχει το λόγο από την ομάδα των σοσιαλιστών είναι εκτός μικροφώνου. Ο κύριος Βουλευτής από τη Μάλτα. Χρειάζεται συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών και η έλλειψη τέτοιων πολιτικών και διαθροτικών, τα διαθροτικά προβλήματα σε ένα κάτω μέλο μπορεί να απειλήσουν σταθερότητα όλων. Εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που οδηγήσει και σε ανάπτυξη και σε νέε και καλύτερε θέσει απασχόληση, κοινωνική δικαιοσύνη επίση για του πολίτε. Τα ωφέλη τέτοιων μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να είναι το καλύτερο κίνητρο αυτό κάθε αυτό για να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσει τουλάχιστον μέσω μακροπρόθεσμα. Η επιτυχής εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι κάτι που θα στερνιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, κυρίω στο επίπεδο στο οποίο οι μεταρρυθμίσεις αυτέ γίνονται αισθητέ. Τα εθνικά κοινοβούλια έχουν βασικό ρόλο για πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων μέσω τη κατάλληλη νομοθεσία, Να μην αναφέρουμε το γεγονό, ότι εμεί είμαστε πιο κοντά στο σημείο όπου γίνονται αισθητά τα αποτελέσματα των αποφάσεων. Στη Μάλτα η πολιτική και από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούν να έχουν στενές σχέσεις και να ακούσουν το εκλογικό σώμα. Όμως πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ εντοπισμού προκλήσεων και αντιστοίχων συστάσεων επιτρέποντας στους εμπλεκομένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνήσεων, στα εθνικά κοινοβούλια και τους κοινωνικούς εταίρους, την ευελιξία την κατάλληλη, να προσεγγίσουν τα προβλήματα με το βέλτιστο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Μια τέτοια ευελιξία στη χρήση δημοσιονομικών μέσων είναι κάτι πολύ βασικό, κρισίμου σημασίας για τη χώρα μας ήταν και κρισίμου σημασία για να φτάσει η χώρα μας εκεί που είμαστε σήμερα. Μια χώρα με ισχυρή σταθερή οικονομία, με υψηλά ποσοστά ανάπτυξης και χαμηλή ανεργία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος. Κύριος Φενιβέζη από την Ουγγαρία, από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ουγγαρία καλωσορίζει το γεγονός ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με αργούς ρυθμούς βγαίνει από την κρίση. Η οικονομική ανάπτυξη είναι ορατή και η ανεργία ε, δείχνει θετικές τάσεις. Η Προεδρία του Συμβουλίου έχει καταβάλει προσπάθειες για τη βελτίωση της καταστάσεως. Η Αυστριακή Προεδρία εξακολουθεί να έχει στη διάθεσή της κάποιους μήνες για να πετύχει κι άλλους στόχους. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και όλη η διαδικασία έχουν βελτιωθεί σαν διαδικασία τα τελευταία δύο χρόνια. Το συζητήσαμε αυτό και στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Το συζητάμε τακτικά στο Κοινοβούλιο και καλούμε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τοποθετηθούν. Μια κοινή κατανόηση του πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι η σωστή προσέγγιση και είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη πραγματικά θα εξετάσουν τις συστάσεις αναχώρα σαν κάτι που βοηθάει και να εφαρμόζουν τις συστάσεις αυτές. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρούσα διαδικασία. Τα μέτρα είναι καλά ως έχουν. Οι συστάσεις αναχώρα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μακροπρόθεσμη στρατηγική, πλήρη στρατηγική και δεν μπορούν να αποτελέσουν μοναδική βάση πολιετούς σχεδιασμού. Η οικονομική ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης έχει επιτευχθεί κυρίως χάρη στην οικονομική σταθερότητα παρόλο που ε, δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σχέση σε τι ατού μεταξύ Ταμείων Συνοχής και μακροοικονομικής πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και σχετική διαδικασία θα αντιμετωπίσουν σοβαρές προκλήσεις μετά τις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο και κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Η καινοτομία, η έρευνα, η ανάπτυξη, η ψηφιοποίηση, όλα αυτά θα αποκτήσουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση, αυτό είναι πρόσδεκτο, αλλά η χρηματοδότηση νέων τομέων δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος παραδοσιακών τομέων της πολιτικής συνοχής και της αγροτικής πολιτικής, διότι αυτά ήταν πολύ σημαντικά εργαλεία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη θέλουν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια εφοδιασμού σε τρόφιμα, καθώς και τη διατήρηση του εργατικού δυναμικού της υπαίθρου που είναι κάτι πολύτιμο για την ευρωπαϊκή οικονομία. Σας ευχαριστώ την προσοχή σας. ευχαριστώ, λέει Δεν έχουμε άλλους ομιλητές. Γνωρίζουμε ότι δεν έχουν λάβει το λόγο όλες οι χώρες που εκπροσωπούνται πριν πω εγώ ίδιος κάτι, ο κύριος Μαυρίδης θα πει κάτι, αλλά έχουμε χρόνο. Κανείς δεν υποχρεούται να ομιλήσει. Αλλά αν κάποιοι από εσά επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη συζήτηση, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να το ζητήσετε. Αναφέρθηκε ότι ήθελα να μιλήσει και ο Παπαδημούλης, ο πρόεδρος λέει δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Όταν καταφθάστηκε θα του δώσουμε το λόγο. Εν τω μεταξύ, πέρα από εκείνον που είναι στον κατάλογο, αλλά δεν είναι παρόν τώρα, εγώ έλεγα κάτι άλλο. Ότι από τα εθνικά κοινοβούλια, από του συναδέλφου των εθνικών κοινοβούλιων, είναι κάποιοι που δεν έλαβαν το λόγο. Και αν επιθυμούν, α το κάνουν. Διότι αρχικά ήμασταν πιο απεσιόδοξοι όσον αφορά τη δυνατότητα να δώσουμε το λόγο σε όλους και ήμασταν πολύ αυστηροί μόνο ένας αναχώρα κλπ. Τώρα υπάρχει χρόνος. Αν το επιθυμείτε ε, μπορείτε να συμμετάσχετε στη συζήτηση. Ίσως ο ίδιος να εκφράσω κάποιες ε, σκέψεις εάν κατά τη διάρκεια της παρεμβάσεώς μου κάποια από εσά αποφασίσετε να λάβετε το λόγο εκ νέου ή να λάβετε το λόγο για πρώτη φορά, θα έχετε δυνατότητα να το επισημάνετε στη γραμματεία. Σημειώνω κάποια σημεία που εφήγησαν. Διεφάνησαν κάποια σημεία από τη συζήτηση. Ιδώθηκαν τα σημεία από διάφορες οπτικές γωνίες. Αυτό δείχνει βέβαια πόσο δύσκολο είναι να ρυθμίσουμε μια κοινή οικονομική διακυβέρνηση σε μια ένωση, σε μια νομισματική ένωση που δεν είναι απόλυτα ολοκληρωμένη και τίθεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να σχολιάσω κάποια από τα σημεία που άκουσα. Ένα σημείο ήταν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Εκεί υπάρχουν δύο ομάδες προβλημάτων. Η μία κατηγορία. Τι είδου οικονομικό πρότυπο οικονομικής διακυβέρνησης προτιμούμε. Δεύτερον, χρειαζόμαστε κάποιους κανόνες ή δεν χρειαζόμαστε κανόνες. Προσωπικά εγώ, όπως γνωρίζετε, είμαι ένθερμος υποστηριχτής του αναγκαίου βαθμού ευελιξίας όσον αφορά ε, το Συμφώνου Σταθερότητας ε, και Ανάπτυξης. Δεν πιστεύω, ότι, δεν πιστεύω ότι είναι τέλειοι αυτοί οι κανόνες, μάλιστα είναι αρκετά ατελείς κατά την άποψή μου, για διάφορους λόγους. Απ' την άλλη βέβαια, και γι' αυτό εξετίμησα την παρέμβαση του κ. Ριμπόλα από το Ιταλικό Κοινοβούλιο, που δεν είναι και το κόμμα μου, είναι το αντίθετο κόμμα στο οποίο ανήκει αν υπάρχει διαφορετικός, διαφορετικό τόνο άκουσα από τους άλλους τόνους ομιλιών που άκουσα. Κανείς δεν αμφισβητεί το ότι υφίστανται κάποιοι κανόνες. Κάποιος μπορεί να πει δεν μου αρέσουν οι κανόνες. Δεν συμφωνώ με τον τρόπο που εφαρμόζονται οι κανόνες. Μπορούμε να αμφισβητήσουμε όμως το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε μετά κατά πόσο αυτοί οι κανόνες είναι σωστά εφαρμοσμένοι και κατά πόσο οι κανόνες αυτοί, αυτοί καθ' αυτοί οι κανόνες είναι ορθοί. Για το πρώτο σημείο, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό, να σχολιάσω την συζήτηση που γίνεται στην Ιταλία περί προϋπολογισμού. Δύσκολο να αμφισβητηθεί το ότι το, το, το, το έγγραφο το οικονομικό δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες. Οι ίδιοι κανόνες χωρίς την ευελιξία που απαιτεί 0,6% σύμφωνα με την περίφημη μήτρα για διαθωτικές μεταρρυθμίσεις και μια μείωση 0,8 επιδείνωση 0,8 προτείνει η κυβέρνηση. Υπάρχει διαφορά 1,4 μεταξύ στόχου και προτάσεως της κυβέρνησης. 1,4 είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντική απόκληση όπως αποκαλείται. Εγώ προτείνω στους Ιταλούς φίλους μου είναι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι αυτό είναι σημαντική απόκληση, δεν μπορείτε να προσβάλλετε τον Επίτροπο, διότι αυτή είναι σημαντική απόκληση. Είναι γεγονό. Είναι στοιχείο, γεγονό. Και στο έγγραφο τη κυβερνήσεω αναφέρεται ω σημαντική απόκληση, διότι είναι σημαντική. Ξέρουμε ότι σύμφωνα με του κανόνε το περιθώριο τη ευελιξία απόκληση είναι μέχρι 0,05 και σε κάποιοι κανόνε ότι σε δύο χρόνια 0,25. Α ξεκινήσουμε από το 0 είναι 0,5 ας πούμε. Από 0,5 και 1,4 ε, υπάρχει 0,9. Ε, Άρα ξεπερνάει κατά πολύ το περιθώριο της ευελιξίας. Πέραν αυτού, ε, καταρχήν, σύμφωνα με τους τρέχοντες κανόνες αυτό δεν γίνεται, ας πούμε ότι μπορείτε να προσθέσετε κάθε ευελιξία που είναι εφικτή. Οπότε η διευθυντική μεταρρύθμιση, ο κανόνα περί μεταρρύθμιση και επενδύσει έχει ένα ανώτατο όριο. Ξανά δεν μπορείτε να φτάσετε στο 1,4. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκληση. Είναι γεγονό. Τι σημαίνει ότι δεν έχει σημαντική απόκληση. Μπαίνει στη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματο. Αν μπει στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο, αυτό δεν στιγματίζει κανένα. Πολλέ χώρε μπήκαν στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο, όπω είναι η Ισπανία τώρα. Κάθε χώρα, νομίζω, εκτό από δύο-τρει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μπήκαν στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο. Δεν μπορούμε να πούμε, αλλά η Γαλλία παραβιάζει το έλλειμμα, παρεύει το, το έλλειμμα. Αν συνέβη, μπαίνει στην διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, αν μπει, μένεις εκεί και λες διασκώ την οικονομική μου πολιτική αν θέλω. Αλλά δεν προσβάλλεις έτσι την, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευάνης σε αυτή τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Αυτοί είναι οι κανόνες. Αν η συζήτηση ήταν πιο μετριοπαθής, όπως υπήρξε στην παρέμβαση του κυρίου Ριμπόλα, θα έχουμε πολύ λιγότερη ένταση στις αγορές. Και αυτά μπορούμε να πούμε θέλουμε την τάδε δίνα ευελιξία. Μπορεί μπορεί να πει κανεί ότι μπορώ να μείνω στο καθεστώ υπερβολικού ελλείμματο για ένα-δύο χρόνια για ανάπτυξη ή θέλω αυτά τα μέτρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά είναι τα σωστά, αλλά θα ήταν μια λογική που θα μπορούσε να ακολουθηθεί αντί να δημιουργήσει κανεί μια συζήτηση και αντιπαράθεση για την ύπαρξη του κανόνα. Ότι θα... και ότι υπάρχει μηχανογραφία κατά κάποιε κυβερνήσεως. Αν παραμείνει συζήτηση σε αυτόν τον τόνο, είναι χρήσιμη συζήτηση. Μπορεί να διεξαχθεί. Και πέραν αυτού, θα σχολιάσω και άλλε παρεμβάσει. Μπορώ να πω ότι πράγματι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε αρκετά εργαλεία για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη, την απασχόληση. Αυτό αληθεύει. Για να τα πω ειλικρινά, κάποιοι από εμά πιστεύουν ότι θα έπρεπε να έχουμε στρατηγική επενδυτική, επενδυτικά εργαλεία, κανόνε περί επενδύσεων, μεγαλύτερο κονδύλι, αν δεν θε συνεχώ να πολεμήσει στα ε, ε, στα επίπεδα εθνικού προπολογισμού να έχει κοινό προπολογισμό ή μετά να έχει πειθαρχία στην αγορά είναι υποχρεώσει σε εθνικό προπολογισμό να συμμορφωθεί. Μα δείχνει η συζήτηση ότι η μόνη λύση πρέπει να βρεθεί. Πρέπει να ολοκληρωθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Να έχει πιο αποτελεσματικά εργαλεία. Οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη θέλουμε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα μιλώ σαν ένα μέλος που παίρνει το λόγο στη συζήτηση. Μετά στην Επιτροπή υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Είναι αυτοί που θέλουν δημοσιονομική υπευθυνότητα, άλλοι ακολουθούν και νησιανή προσέγγιση. Είναι και οι δύο συμβατέ προσεγγίσεις. Και μετά η δημοκρατία, αλλά με τι εκλογές, επιλέγει την κυβερνητική πολιτική τη δέωσα μπορεί να επικρατήσει και υπάρχει εθνικό κομμάτι και ευρωπαϊκό κομμάτι όπου εκεί παίζουν ρόλο και ευρωπαϊκέ εκλογέ για να καθορίσουν τη λύση. Είχαμε περισσότερο συντηρητική Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προηγούμενη θητεία και πιο αυστηρή εφαρμογή δημοσιονομικού συμφώνου σταθερότητα. Και τώρα είχαμε περισσότερο κεντροαριστερή Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό είναι λογικό. Και ο πολίτη μπορεί να αποφασίσει. Μπορεί να έχει διαφορετική εντύπωση και, και απόψεις. Αυτό που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου, σας εκφράζω, και η συζήτηση που γίνεται μεταξύ μελών του Ευρωκοινοβουλίου και μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου, η συζήτηση γίνεται επικοδομητικά και βοηθά να γεφυρώσουμε διαφορές οπτικών γωνιών, επικότητα, εθνικότητα. χωρίς, χωρίς να αγνοούμε τις υγιείς διαφορές που υπάρχουν σε μια ένωση των 27. 28 σημαίνει στο μέλλον 27 με πολλά εκατομμύρια πολίτες. Διαφορές λοιπόν που είναι υγιείς. Μπορούν να συμβιώσουν χωρίς να αμφισβητήσουμε την, ύπαρξη της, την ίδια τη συνύπαρξη. Λοιπόν, καλωσορίζω την επικοδομητική συζήτηση που έγινε. Λοιπόν, οι δημοσιονομικοί κανόνε του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη δεν αφορούν το έλλειμμα και το χρέο, αλλά και η μακροοικονομική σταθερότητα και ανισορροπίε. Αυτό το κομμάτι του συμφώνου εφαρμόστηκε λιγότερο από το άλλο. Το είπε και η Περβάνς. Και το μέλος τη Λέγκα του Βορρά. Λέγατε παρόμοια πράγματα. Βλέπετε πώ αυτή η συζήτηση μπορεί να παράσχει πολύ διαφορετικού συνδυασμού θέσεων. Χρησιμότατο. Πολύ ενδιαφέρον και η Ιταλία επίσης είναι κοντά στη διαδικασία υπερβολικού χρελήματος. Αν ρωτάτε ένα Ιταλό τι θέλει, τελικά αν θέλει να ισχύσει, να ισχύσει αυτό, είναι σαν να αυτοπυροβολείστε κάπως, να αυτομολοπίζεστε. η εμπορική θέση, αυτό πάνω από 6% που θέλετε να βάλετε, είναι κάτι που παραβιάζει τον κανόνα που, που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χώρα. Που έχει... Δεν είναι ότι δεν συμβαίνει κάτι. Λοιπόν, καμιά φορά δεν ακούμε ένα τον άλλον, γιατί διατείνονται ότι άλλα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα θέμα είναι αυτό. Κάτι άλλο που θεωρώ άκρο ενδιαφέρον στα σχόλια που άκουσα. Μακροοικονομική ρεσιμότητα στενή διασύνδεση μεταξύ οικονομικής πολιτικής, δημοσιονομικής εποπτείας και συμφώνου σταθερότητας και χρήσεως των χρημάτων συνοχής. Εδώ είμαστε διχασμένοι στο Κοινοβούλιο. Το καταλαβαίνω ότι σε εθνικά κοινοβούλια δεν ενδιαφέρεστε πολύ γι' αυτό. Είναι χρήσιμο λοιπόν να συνομιλήσετε με την κυβέρνησή σας, γιατί το θέμα τώρα είναι θέμα συζήτησης στον κανονισμό που θα διέπει τη νέα φάση των ιδιωτικών ταμείων και κατά πόσο θα, είναι, θα υπάρχει μακροοικονομική αιρεσιμότητα, οι ρεσιμότητες θα έχουν σήμερα, που ποτέ δεν εφαρμόστηκαν και προσπάθησαν να εφαρμοστούν στην Πορτογαλία και την Ισπανία και ο κόσμος τελικά είπε όχι, δεν γίνεται. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ήταν χρήσιμο να συζητηθεί στα εθνικά κοινοβούλια. Να συνομιλήσουν τα εθνικά κοινοβούλια με την κυβέρνησή του, γιατί αυτό θα ενταχθεί στον τριμερή διάλογο πολύ σύντομα. Και εμεί το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, απλώ διάλεξα κάποια ενδιαφέροντα θέματα που συζητήθηκαν. Βλέπω ότι ο κ. Παπαδημούλης κατέφθασε, οπότε μπορώ να σταματήσω που προσπαθούσα να σε διασκεδάσω και να κερδίσω χρόνο. Μπορώ να σταματήσω τώρα. Βέβαια, έχουμε μέχρι τις 4.30. Από την εμπειρία μου, Λοιπόν, έχουμε μεγαλύτερη, είχαμε μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα που κάναμε το Φεβρουάριο και πάντα το τον να Έχουμε πρώτο τμήμα όπου όλοι προετοιμάζουν ομιλία. Και αυτό είναι πολύ καλό. Το καλύτερο κομμάτι είναι το τελευταίο κομμάτι. Όπου αρχίζουμε την πραγματική διάδραση και μιλάμε και κουβεντιάζουμε και απαντάμε ένα στον άλλο. Αυτό το καλύτερο κομμάτι και το χρησιμότερο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα χρησιμοποιήσουμε το τελευταίο μισάωρο άριστα σε αυτό το πνεύμα, πιο ελεύθερη συζήτηση, κουβέντα μεταξύ μα. Δημήτρη, πρώτα εσύ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη γιατί ήρθα ασθμένον πάλι στην αίθουσα, αλλά την ίδια ώρα είχαμε και μια άλλη επιτροπή όπου έπρεπε να με παρών. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι συμμερίζομαι πολλές από τις εισαγωγικές παρατηρήσεις του εισηγητή μας, του κυρίου Κώστα Μαυρίδη, που είχε την ευκαιρία να ακούσω ε, στην αρχή η βασική μου παρατήρηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η Ευρωζώνη δεν κάνει τα βήματα που είναι απαραίτητα για να προετοιμάσει τον εαυτό της και τα κράτη-μέλη απέναντι στη νέα κρίση που κάποια στιγμή θα έρθει γιατί η κρίση κάνει κύκλους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Τραπεζική Ένωση. Προχώρησαν οι δύο πυλώνες, αλλά ο τρίτος πυλώνας, που είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων, έχει παραπεμφθεί στις αρχές ελληνικές καλένδες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέλει, η Κομισιόν το έχει προτείνει, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει για να μην κινδυνεύσουμε από νέες συστημικές κρίσεις, αλλά το θέμα έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο, όπου κάποια κράτη-μέλη ουσιαστικά βάζουν φρένο, έχουν ένα άτυπο βέτο. Ένα δεύτερο θέμα είναι ο περιορισμός της τεράστιας φοροδιαφυγής μέσω των tax rulings. Πριν από λίγες ώρες ήταν εδώ η Επίτροπος Ανταγωνισμού, η κυρία Βεστάγκερ, η οποία μας έλεγε ότι με νόμιμο σε πολλά εισαγωγικά τρόπο πάρα πολλές πολυεθνικές καταφέρουν να μην πληρώνουν καθόλου φόρο για τα τεράστια υπερκέρδη τους γιατί κάποια κράτη-μέλη έχουν βρει ένα νόμιμο τρόπο να τις απαλλάσσουν από τη φορολογία. Και αυτό επιβαρύνει με υπερφορολόγηση τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εμποδίζει έναν υγιή επιχειρηματικό ανταγωνισμό υπέρ των γιγάντων και σε βάρος των αδυνάτων. Ένα, ένας τρίτος τομέας είναι η φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, όπου καθυστερεί η εξέβρεση κανόνων έτσι ώστε οι γίγαντες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης να συμβάλλουν και αυτοί στα φορολογικά έσοδα. Οι περιπτώσεις της McDonald's στην στο Λουξεμβούργο για το tax rulings είναι ένα παράδειγμα, η περίπτωση της Google είναι ένα άλλο παράδειγμα. Κλείνοντας, για να μην μιλήσω πολύ, θα ήθελα να πω ότι είμαι ικανοποιημένος γιατί μετά από τέσσερα περίπου χρόνια θητείας αυτού του Ευρωκοινοβουλίου η χώρα μου η Ελλάδα έχει εξέλθει πια από τα μνημόνια και έχει μπει στον κανόνα της ε, παρακολούθησης της συζήτησης της εποπτείας για το πώς ακολουθούνται και εφαρμόζονται οι κρατικοί προϋπολογισμοί μέσω της Κομισιόν μέσα από τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού ε, Εξαμήνου. Και θεωρώ ε, αναγκαίο να υπογραμμίσω σε μια περίοδο που στη γειτονική Ιταλία σημειώνονται αρκετές αναταράξεις ότι σε αντίθεση με την γειτονική μας Ιταλία η Ελλάδα έχει καταφέρει να έχει όχι δημοσιονομικά ελλείμματα αλλά δημοσιονομικά πλεονάσματα και έχει μπει σε μια πορεία σταθερής ανάκαμψης της οικονομίας μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια στην Ελλάδα επίσης. Οπότε, είχα κάνει... Είχα και εγώ ένα ερώτημα που θα μπορούσα να απαντήσεις, Δημήτρη, για το θέμα του νέου προϋπολογισμού και τη θέση σε σχέση με τις συντάξεις. Αυτό το, τις περικοπές των συντάξεων. Θέλεις να μιλήσεις? Πρώτα ο συνάδελφος και μετά εσύ. Πέρα το συνάδελφό σου. Ο κύριος Μπαλούρας. Κύριε Πρόεδρε, ε, θέλω να σημειώσω τις κρίσιμες ε, διαπιστώσεις που κάνατε, οι οποίες είναι προωθητικές για ένα διάλογο σε βάθος. Πρέπει να φύγουν οι, τα, τα στημένα ε, φοβικά σύνδρομα που υπάρχουν από πολλές πλευρές στην Ευρώπη. Ε, θυμίζω τώρα για το θέμα που θίξατε ε, και ευχαριστώ που το θίξατε. Θα μιλήσει και ο Αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Παδημούλης, ε, ξέρετε ότι η περικοπή των συντάξεων επιβλήθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ε, το οποίο δογματικά για μία ακόμα φορά έτσι, έκανε λάθος στις προβλέψεις του. Είχε κάνει επανειλημμένα λάθος, θυμόσαστε τον πολλαπλασιαστές που βγαίνανε έξω και όλα αυτά. Λοιπόν, επέβαλε αυτή την περικοπή των συντάξεων λέγοντας ότι δεν θα πιάσουμε ούτε τα πρωτογενή πλεονάσματα ούτε την ανάπτυξη. Τώρα έχουμε πιάσει επί τρία συνεχή χρόνια υπερπλεονάσματα ξεπερνώντας το 3,5% το οποίο είναι πάρα πολύ αλλά τα έχουμε πιάσει και δεύτερον έχουμε ανάπτυξη αρκετά δυναμική. Φέτος θα έχουμε δύο και κάτι και του χρόνου, όπως είπε προχτές μάλιστα το Δουνουτού, με νέες προβλέψεις θα έχουμε 2,5%. Ε, ε, θέλω να πω όμως ένα στοιχείο για την περικοπή των συντάξεων. Οι συνταξιούχοι, ε, κύριε Πρόεδρε, στην Ελλάδα και προφανώς και στην Ιταλία, ε, δεν είναι, επειδή είναι βαθιά η κρίση και όπως ανέφερα και στην πρωτομιλία μου, οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές, ενισχύουν οι συνταξιούχοι έτσι, τους ανέργους, τα παιδιά τους που είναι άνεργα ή ζουν με ανέχεια, τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους. Επομένως αυτό θα είναι ένα εισόδημα που θα διαχεθεί, αν θέλετε να μιλήσουμε και τις επιπτώσεις στην οικονομία, θα διαχεθεί στην οικονομία. Έτσι ώστε να, να, να ενισχύσει και την ανάπτυξη και τα άλλα στοιχεία της ανάκαψης που χρειαζόμαστε. Ε, θέλω να σημειώσω, να σημειώσω επίσης εδώ και τελειώνω ότι θα πρέπει να είναι καθαρή η απόφαση και των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και του Διεθνούς Νοσματικού Ταμείου γιατί οποιαδήποτε σκιά να φεθεί τότε οι αγορές θα το εκμεταλλευτούν και είμαστε μπροστά στην έξοδό μας σε αγορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρέμβασή σας και, το, και το λόγο που μου δώσατε. Δημήτριος, please. Ε, ναι, είμαστε στην Ελλάδα αισιόδοξοι ότι μπορούμε να πετύχουμε τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα και να τις στηρίσουμε απολύτως και για το 2018 και για το 2019. Η χώρα μου, η Ελλάδα, έχει δεσμευτεί ότι θα πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% και το 2018 και το 2019. Για το 2018 που πλησιάζουμε προς το τέλος της χρονιάς, οι εκτιμήσεις της Κομισιόν είναι ότι όχι μόνο θα το πιάσουμε, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Οι εκτιμήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων της Κομισιόν και του ESM μιλούν για πρωτογενές πλεόνασμα που θα ξεπεράσει και το 4%. Πέρσι ξεπέρασε και πάλι το 4%, ήταν 4,2%, ενώ η δέσμευση ήταν 1,75%. Και τώρα η επιδίωξή μας είναι να πείσουμε τους πάντες και την Κομισιόν και τον ESM και το Eurogroup, ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι πάκτα σουν σερβάντα, θα πετύχουμε το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% και το 2019, χωρίς το αχρίαστο και αντιαναπτυξιακό μέτρο της περικοπής των συντάξεων, της πρόσθετης περικοπής των συντάξεων, γιατί οι συντάξεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου 40%. Και επειδή όλοι εκπροσωπείτε πολίτες, θα ήθελα να αναρωτηθείτε αν θα ήταν εύκολο στη χώρα κάποιος τη δική του να κόψει τη σύνταξη κατά 40%. Ο στόχος μας όμως είναι να πιστούν όλοι με βάση τους αριθμούς και προς τα εκεί κινούμαστε γιατί μόλις χτες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διόρθωσε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ενώ τον Απρίλιο που έβλεπε για το 2019 ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 1,8%, οι χθεσινές ανακοινώσεις και προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μιλούν για 2,4%. Τι συνέβη στην Ελλάδα δηλαδή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με καθυστέρηση πολλών χρόνων που έκανε απεσιόδοξε προβλέψει ήρθε να συμφωνήσει με αυτά που προέβλεπε η Κομισιόν και η ελληνική κυβέρνηση εδώ και χρόνια. Το μέτρο αυτό επιβλήθηκε από, τον, από την αιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στηριγμένο σε προβλέψεις που δεν επιβεβαιώθηκαν. Δεν το ζήτησε ούτε η Κομισιόν, ούτε ο ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε το Eurogroup. Και πριν μία εβδομάδα έγινε Eurogroup όπου οι πάντες και ο πρόεδρος του Eurogroup ο κύριος Σεντένο και ο αρμόδιος επίτροπος ο κύριος Μοσκοβισή και ο κύριος Ρέκλινγκ, ο επικεφαλής του ESM, μίλησαν με θετικά λόγια για την πορεία υλοποίησης των ε, δημοσιονομικών στόχων της Ελλάδας και τώρα που είμαστε εκτός μνημονίου, οι δεσμεύσεις μας ισχύουν 100% αλλά είναι ευθύνη της χώρας της κυβέρνησής της, του κοινοβουλίου της, να επιλέξει το μείγμα πολιτικής με το οποίο θα πετύχουμε τους στόχους. Επομένως, τηρούμε 100% τους στόχους, αλλά περιμένω από τους κοινοβουλευτικούς των άλλων κρατών μελών να σεβαστούν και το δικό μας δικαίωμα να αποφασίζει το κοινοβούλιο μας όπως αποφασίζει και το δικό σας κοινοβούλιο για το πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά και ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, ο πρόεδρος της ΕΚΟΝ, που έχει ασχοληθεί και πολύ με την Ελλάδα, έχει διαπιστώσει ότι όσα σας λέω είναι απολύτως ακριβή και στηρίζονται στους αριθμούς. Thank Σας ευχαριστώ. η Ελλάδα έχει μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα και έτσι βγήκε από την διαδικασία υπερβολικού χρέου για αυτόν τον λόγο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τώρα η Ελλάδα ξεπερνάει τον όρο του πρωτογενούς πλεονάσματος και του ελλείμματος. Το συμπληρωματικό 1% που είχε προβλεφθεί αρχικά από το δούνο του επετεύθη βάσει προβλέψεων που δεν υλοποιήθηκαν. Και τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά, αλλά είναι πολύ λογικό αυτό. Σοφή απόφαση να γίνει αυτή η αλλαγή στον προϋπολογισμό. Ο κύριος Αβέροφ Νεοφίτου, πρόεδρος της Μόνης Επιτροπής για Δημοσιονομικά Θέματα και Προϋπολογισμού της Κύπρου από το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Όντως και η Ελλάδα κατάφερε να βγει από τα μνημόνια με μια πορεία με προβλήματα και στον λαό και στους πολίτες που διάρκησαν 8 χρόνια. Όμως ε, βρίσκεται σήμερα ε, στην πορεία της οικονομικής ανάπτυξης και όπως είπε ο συνάδελφος και πέραν των ε, εκτιμήσεων και των προβλέψεων. Θα μπορούσε κάλλιστα και η Ελλάδα να είχε μειώσει τα προβλήματα αντί 8 χρόνια θα μπορούσε και η Ελλάδα στα 3-4 χρόνια να είχε βγει από τα μνημόνια. Ε, και είναι και μια απάντηση αυτή σε όσους θεωρούν τα μνημόνια ως κατάρα. Μας δίνουν την ευκαιρία να διορθωνόμαστε. Και έχουμε μόνο επίσης τα παραδείγματα της Ιρλανδίας, τα παραδείγματα της Πορτογαλίας, της Κύπρου και τώρα της Ελλάδος. Με μια επιφύλαξη όμως, για να μην ξαναοδηγούμε τις χώρες μας σε δημοσιονομικές περιπέτειες. Πρέπει να έχουμε ένα κανόνα υπόψη μας. Τα έσοδα δεν είναι πάντα σταθερά. Όταν όμως αυξάνεις τις ανελαστικές δαπάνες, αυτές παραμένουν μόνιμες. Και σε περίπτωση μια έστω και μικρής ύφεσης ή χαμηλότερου ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, η δημοσιονομική εκτροχίενση θα είναι μπροστά σου και πάλι θα οδηγήσει τη χώρα σου σε περιπέτειες. Και εμείς στην Κύπρο αναγκαστήκαμε και μισθούς και συντάξεις όχι στα επίπεδα της Ελλάδος να το πράξουμε. Όμως ήταν αναγκαίο να το πράξουμε για να μπορούμε να δίδουμε έστω και μειωμένε συντάξεις και μειωμένους μισθούς. Εάν δεν το κάναμε αυτό δεν θα μπορούσαμε να δίδουμε καθόλου συντάξεις και καθόλου μισθούς. Με αυτή την προσέγγιση θεωρώ ότι αν γίνει χτήμα όλων μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πιο σταθερές συνθήκες και για την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και για τις χώρες μας. Ένα τελευταίο. Και η Ελλάδα και η Κύπρος και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία πληρώσαμε και μέρος του κόστους των ελλημάτων των ευρωπαϊκών πολιτικών. Μπήκαμε στη ζώνη του ευρώ. Εισάξαμε το ευρώ ως νόμισμά μας έχοντας μόνο ως ενιαία πολιτική την νομισματική. Και για χρόνια είχαμε 16 και 17 διαφορετικές νομισματικές πολιτικές. Τώρα με το Six Pact και τις άλλες πρωτοβουλίες που λήφθηκαν μπαίνει μια τάξη και όσον αφορά το δημοσιονομικό σκέλος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρκετά περίπλοκοι κανόνες μας. Συμφωνώ όμως ότι θέλαμε να ευθυγραμμίσουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αν δεν έχουμε άλλους ομιλητές, ήρθε η ώρα ο εισηγητής μας να λάβει το λόγο. Κύριε Μαυρίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μητρική μου γλώσσα. Ε, έχω ακούσει με προσοχή όσα έχουν λεχθεί σήμερα. Υπάρχουν θέματα που δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε Υπάρχουν όμως θέματα για τα οποία θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε μια σύγκληση και θα επικεντρωθώ σε αυτά. Για παράδειγμα, εάν κάποιος επιμένει ότι με το να μειώνει τη φορολογία στους πλούσιους και ταυτοχρόνως να παρέχει κοινωνικές δαπάνες, αυτό είναι σοφή και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, δεν θα μας βρει ποτέ σύμφωνος. Όμως θα επικεντρωθώ πολύ σύντομα σε δύο-τρία σημεία που νομίζω ότι <clears throat> πρέπει να υπάρξει ευρύτερη συνένεση. Ακούγοντας την περίπτωση της Ελλάδας, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό επιχείρημα η ανάγκη για flexibility στα European Rules δεν είναι το flexibility in European rules, δεν είναι για ούτως ώστε κάθε κράτος μέλος να κάνει ό,τι κόψει του κεφαλιού του. Είναι γιατί όπως το ακούσαμε, εάν υπήρχε flexibility και ιδιαίτερα αν είχαμε τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, το τεράστιο ζήτημα που λέγεται ανθρώπινη δυστυχία θα ήταν σαφώς μειωμένο. Και αν έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας, αυτό νομίζω πρέπει να το δείχνουμε στην πράξη στις δύσκολες ώρες. Τελειώνω με το εξής. Για όσους θεωρούν ότι η Επιτροπή είναι σωστή, θα πω ότι και η Επιτροπή το 2015 εισηγήθηκε ευελιξία στους κανόνες αυτούς, αλλά θα πω επίσης ότι πολλές φορές η Επιτροπή ναι λειτουργεί αντίθετα από την κοινή λογική και αντίθετα από την αλληλεγγύη μεταξύ μας. Θα μείνω μόνο σε ένα σημείο. Cohesion funds and cohesion policies. Πώς είναι δυνατόν να πείσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες ότι απαιτούνται μακροοικονομικές προϋποθέσεις για ένα κράτος μέλος, ούτως ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτού του είδους τα ταμεία αυτά τα ταμεία έγιναν ούτω ώστε να έχουμε κοινωνική συνοχή. Το να θέτουμε προϋποθέσεις, προϋποθέσεις με συγχωρείτε, είναι ουσιαστικά τιμωρία στα κρατη για να έχουν πρόσβαση τη στιγμή που τα έχουν ανάγκη. Γι' αυτό και η θέση της ομάδας μου είναι ξεκάθαρη σε αυτό το σημείο. Κλείνω, Πρόεδρε, με μια τελευταία κουβέντα. Όποτε ακούσω κάποιον να μιλάει for deepening the EMU, θα περίμενα αυτός ο άνθρωπος να λέει ότι χρειαζόμαστε και ευρωπαϊκό σύστημα εγγυήσεως καταθέσεων. Διαφορετικά δεν έχει καθόλου νόημα να μιλάμε για Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και να μην έχουμε μια ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ήταν πολύ ζωντανή, πολύ χρήσιμη η συζήτηση. Το τελευταίο σημείο σας, του συγητού, το ενστερνίζομαι. Η ευελιξία είναι κάτι, η αμφισβήτηση των ίδιων των κανόνων είναι κάτι διαφορετικό και είναι κάτι ασύμβατο με την Ένωση, αλλά Πολλά πρέπει να γίνουν, ούτω ώστε να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση και το σχετικό πλαίσιο ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη διεξαγωγή της συζητήσεω στους επόμενους μήνες και την επόμενη θητεία και ελπίζουμε ότι το κοινό πλαίσιο αυτών των συζητήσεων και στα Εθνικά Κοινοβούλια θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αμφιβολίες, φόβους και αντίστοιχη έλλειψη εμπιστοσύνη. Σα ευχαριστώ εκ νέου, σα ευχαριστώ όλου και πάμε στο επόμενο σημείο. Α, όχι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών και μετά θα ξεκινήσουμε με το επόμενο σημείο. Πρέπει να γίνει μια ανακατάταξη, αναδιάταξη τη αίθουσα. Αν οι φίλοι μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια επιθυμούν να παραμείνουν, είστε ευπρόσδεκτοι, άκρο ευπρόσδεκτοι, να παρακολουθήσετε τη συζήτηση επί του επόμενου σημείου και την ημερήσια διάταξη. Το επόμενο σημείο είναι πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συμπεριλαμβάνει κάποιες διατάξεις του, του φορολογικού συμφώνου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν είναι κάτι πολύ απόμακρο από τα θέματα που συζητήσαμε. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Είναι ανοιχτέ λοιπόν οι πόρτε μα και είσαστε πολύ ευπρόσδεκτοι να παραμείνετε και να παρακολουθήσετε τη συζήτηση. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή πέντε λεπτών.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 Adiós.

Um, λοιπόν, το επόμενο θέμα, το σημείο 19, ενίσχυση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και την ε, μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική κατεύθυνση των κρατών μελών, πρόταση οδηγίας, όπως γνωρίζετε. Πού στοχεύει στην ε, ένταξη στο νέο νομικό πλαίσιο ενός τμήματος του λεγόμενου Δημοσιονομικού Συμφώνου είναι ένα ευαίσθητο και επίμεχο θέμα και γι' αυτό το Συμβούλιο δεν το εξετάζει σε αυτή τη φάση καθόλου. Αλλά πρέπει. Είναι αναγκαίο. Πού είναι ο συγητής. Α, πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε. Ο συγητής είναι η κυρία Χούμπνερ που εκπροσωπείται από τον Μάρκους Φέρμπερ, στον οποίο και δεν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευτυχώς η Τανούτα μου προετοίμασε ένα ωραίο σημείωμα το οποίο θα διαβάσω. Η πρόταση μεταφέρει στην ε, ενωσιακή νομική τάξη την ουσία της, ε, του Συμφώνου του 2013 για την σταθερότητα στην ε, Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ένωση. Είναι μια διακυβερνητική συμφωνία αυτή η πρόταση βασίζεται το άρθρο 16 ε, αυτής της σύμβασης που λέει ότι πρέπει να μεταφερθεί στην ενωσιακή ένωμη τάξη εντός πενταετίας. Η πρόταση ναι. μεταφέρει το μεγαλύτερο τμήμα του άρθρου 3. Δηλαδή η απέτηση τα κράτη-μέλη να έχουν ένα πλαίσιο δεσμευτικής και ε, δεσμευτικών και αριθμητικών δημοσιονομικών κανόνων και να δημιουργήσουν και έναν ε, διορθωτικό μηχανισμό αν υπάρξει ουσιώδης απόκληση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους. Καλωσορίζει την πρόταση αυτή καταρχήν και θεωρεί ότι είναι πολύ θετικό ότι η Επιτροπή θέλει να μεταφέρει αυτή τη συμφωνία. Στο ενωσιακό δίκαιο πρέπει οι διακυβερνητικές ε, ρυθμίσεις να ενταχθούν στην ενωσιακή μέθοδο αλλά θεωρεί ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί σε ορισμένα θέματα. Η έκθεσή τη ασχολείται με τα τέσσερα θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την νομική βάση τη πρόταση. Η Κομισιόν προτείνει τη δεύτερη υποπαράγραφο του άρθρου 126. 14 της συνθήκης που επιτρέπει το πρωτόκολλο 12 που είναι παράρτημα της ε, συμφωνίας αυτής για το, για το υπερβολικό έλλειμμα. Η Κομισιόν ε, το προτείνει γιατί χρησιμοποιήθηκε και για ένα τμήμα ε, ενός κανονισμού του 2011 που ήταν τμήμα του Six Pack. Τότε είχε υποθεί ότι αυτή η δεύτερος ε, υποπαράγραφος επέτρεπε να γίνουν και λιγότερο από το να αντικατασταθεί το πρωτόκολλο. Η οδηγία λοιπόν θέλει απλώς να διευκρινίσει το υπάρχον πλαίσιο. Είναι καθαρά διαδικαστική. Δεν θέλει κατά κανένα τρόπο να αντικαταστήσει το πρωτόκολλο 12. Στο άρθρο 126-14 της συνθήκης υπάρχει και μια τρίτη υποπαράγραφος που επιτρέπει να υπάρξουν αναλυτικοί κανόνες για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου 12. Αυτό θα ήταν ίσως ε, πιο σκόπιμη νομική βάση. Αυτό είναι αυτό που προτείνει και η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Ξέρει όμως ότι το Συμβούλιο επίσης προτείνει να αλλάξει νομική βάση. Η ΑΦΚΟ, που την ξέρει πολύ καλά, η Ντανούτα, στο σχέδιο γνωμοδότησής της συστήνει να γίνει αυτή η αλλαγή. Εάν περάσουμε στην τρίτη υποπαράγραφο, δεν τροποποιούμε το πεδίο εφαρμογή ή το περιεχόμενο της πρότασης. Δεν αλλάζει τη διαδικασία για την έγκριση του κειμένου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Που δυστυχώ παραμένει η διαδικασία διαβούλευση. Αλλά θα αλλάξει τη διαδικασία για την έγκριση του κειμένου στο Συμβούλιο. Η δεύτερη υποπαράγραφο απαιτεί ομοφωνία. Ενώ η τρίτη υποπαράγραφο μόνο ειδική πλειοψηφία. Γι' αυτό αποφάσισε να προτείνει να αλλάξει η νομική βάση. Με στόχο και ελπίζοντας η συμφωνία για αυτό το σημαντικό θέμα να διευκολυνθεί. Δεύτερο θέμα. Αριθμητικά, ε, αριθμητικές τιμές αναφοράς για το έλλειμμα. Η πρόταση της Κομισιόν δεν περιλαμβάνει τέτοιες τιμές αναφοράς. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει. Οι, οι αριθμητικές τιμές, αναφοράς υπάρχουν στο 2 και στην Συμφωνία γενικότερα, όσο δεν καταργείται με αυτή την ε, προσέγγιση υπάρχει περισσότερη ευελιξία που θεωρεί ότι είναι αναγκαία για να σεβαστούμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτή η συμφωνία έχει εφαρμοστεί και ο στόχος της πρότασης είναι οι κανόνες αυτοί να περάσουν από μία ένωμη τάξη, το διεθνές δίκαιο, να περάσουν σε μία άλλη ένωμη τάξη, το ενωσιακό δίκαιο, χωρίς να αλλάξει η ουσία τους. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν με τρόπο που να πει να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο έχουν ε, μεταφερθεί σε εθνικό δίκαιο αυτοί οι κανόνες και εφαρμοστεί. Η μη συμπερίληψη αριθμητικών τιμών αναφοράς συνάδει με αυτό το στόχο. Έτσι θα μπορέσει να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό για όλους τους στόχους, για όλες τις περιπτώσεις και δεν θα έχουμε αναστατώσεις ή απροθυμία εφαρμογής. Χωρίς αυτές τις τιμές αναφοράς η οδηγία δεν χρειάζεται αναθεώρηση στο μέλλον εάν αλλάξουν ε, οι τιμές αναφοράς που αναφέρονται στη συμφωνία γενικότερα και στο ΤΟΥΠΑΚ. Επίσης προτείνει να υπάρξει ένας ορισμός για το τι σημαίνει ουσιώδης απόκληση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους. Είναι πολύ σημαντικό για να πυροδοτείται ο αυτόματος διορθωτικός μηχανισμός. Και δεύτερον, τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κανόνες παρακολούθησης της εφαρμογής των διατάξεων αυτών. Όμως αυτό υπάρχει ήδη για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Γι' αυτό προτείνει να διευκρινιστεί το σημείο αυτό. Όταν ένα κράτος μέλος έχει ήδη δημιουργήσει στα πλαίσια του TUPAC ε, έναν ανεξάρτητο μηχανισμό ελέγχου, μπορεί να επιφορεστεί αυτός ο μηχανισμός και για την εφαρμογή όσων προβλέπει η οδηγία. Προσβλέπει στη συνεργασία με τους κοιόδης και στην πρόθεση αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι η συζήτηση θα είναι έντονη. Και εγώ θα εκφράσω την άποψή μου αργότερα για αυτό το θέμα. Επόμενος ομιλητής, Ιουκ Μπαγιέ, εκλοράς του οποίου υπερβάνουν μέρές. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τον Νίκ Μπαγιέ και ίσως αναφέρω και κάνα δύο σημεία δικά μου ως συντονίστριας. Τι λέει λοιπόν ο Νίκ Μπαγιέ. Μετά την οικονομική κρίση που έχουμε από το 2008 η Ένωση έλαβε δημοσιονομικά μέτρα δραστικά για να υπάρξει πιο στενή επίβλεψη των εθνικών προϋπολογισμών και να είναι πιο ρωμαλαίο το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, γιατί η κατάσταση όπως έχει μέχρι τώρα έχει συμβάλει στην ύφεση. ω Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρεί ότι δεν είμαστε υπέρ του να ενταχθεί αυτή η συμφωνία στις συνθήκες εάν δεν τροποποιηθεί εκ βάθρων αυτή η συμφωνία. Και όπως λέμε μόνιμα από την αρχή αυτής της συζήτησης θα πρέπει να γίνει και μια αξιολόγηση για τις επιπτώσεις αυτού του συμφώνου. Κατά τη γνώμη μας, το TSG πρέπει να αντικατασταθεί από μια συνθήκη που να ενθαρρύνει την οικονομική και κοινωνική σύγκληση των κρατών μελών και ιδιαίτερα των κρατών μελών της Ευρωζώνης, αποφεύγοντας προφανώς να παραληφθούν μέτρα που συνέβαλαν στην όξυνση της λιτότητας. Η Κομισιόν αναλύει μόνο τα δημοσιονομικά δεδομένα. Δεν υπάρχει μια σφαιρική προσέγγιση της οικονομικής κατάστασης της ζώνης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη όλους τους δείκτες, είτε είναι κοινωνικοί, είτε κοινωνικοί, είτε περιβαλλοντικοί και όχι μόνο δημοσιονομικοί Πριν καθορίσουμε τη στάση των κρατών μελών της Ευρωζώνης, γιατί μια σειρά των δεδομένων και των διατάξεων αυτή τη συμφωνία, δεν επιτρέπουν τις επενδύσεις στα κράτη-μέλη. Οπότε δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη, άρα και περισσότερη απασχόληση και επιδεινώνεται η επισφάλεια. Πρέπει λοιπόν να γίνουν αυτά τα πράγματα για να δημιουργηθεί απασχόληση, θέσεις ποιοτικέ εργασίες και για να καταπολεμήσουμε την αυξανόμενη επισφάλεια και ανέχεια. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι ο προπολογισμό είναι αποκομμένο από την καθημερινή ζωή. Αυτό δημιουργεί απαράδεκτε ανισότητες και δεν προωθεί Η λιτότητα που προκάλεσε αυτή η συμφωνία κατακαιρμάτισε την κοινωνία μας. Αυξήθηκε η φτώχεια και μειώθηκε η κοινωνική προστασία. Επειδή υπάρχει όλο και περισσότερη δυσπιστία των πολιτών και επειδή υπάρχει άνοδος των λαϊκισμών, χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να προστατεύει και όχι να ενισχύσουμε τις συνθήκες που ήδη έχουν κάνει πολλές ζημιές για το θέμα της νομικής βάσης. και τις προτάσεις της συζητρίας μας. Ας θυμηθούμε πώς ξεκίνησε αυτό το θέμα. Αυτή η συμφωνία TSCG, όπως λέει και ο Ιγμπαγέ, δεν μπορεί να ενταχθεί στην ενωσιακή νομική τάξη χωρίς να τροποποιηθεί, πρώτα απ' όλα να αξιολογηθεί η λειτουργία της μέχρι τούδε και μετά να διορθωθεί. Ζητήσαμε και την γνώμη ως συντονιστέ της νομικής υπηρεσίας θεωρώντας ότι αν η συμφωνία αυτή ενταχθεί στην ενωσιακή ένωμη τάξη θα είχαμε σύγκρουση των νομικών βάσεων. Από τη μία θα είχε μία νομική βάση αυτή η συμφωνία και από την άλλη, άλλη το six pack και το two pack. Η νομική υπηρεσία όμως προτίμησε να προτείνει άλλη νομική βάση που για μας είναι απόλυτα παράδεκτο. Να περάσουμε από την ομοφωνία στο Συμβούλιο σε μια νομική βάση που απαιτείται μόνο η δική πλειοψηφία. Ενώ αυτή η συμφωνία τροποποιεί θεμελιωδώς το σύνολο των κανόνων που υφίστανται. Δηλαδή το πνεύμα της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 126-14 που θεωρούμε ότι υπάρχουσα είναι η σωστή νομική βάση. Οπότε δεν στηρίζουμε τις προτάσεις Τη συζητήτρια. Ευχαριστώ. λουν συνάδελφε Λούνς από το ECR, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητά συγγνώμη ο που δεν μπορεί να παρασταθεί σήμερα, να παραστεί λόγω των εκλογών της περασμένης εβδομάδας στη Λετωνία και μου ζήτησε να διαβάσω τι απόψει του. Ο Ρόμπερτ Σίλερ σημειώνει την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο πιστεύει ότι ορθά δημοσιονομικά, υγιή, δημοσιονομικά σημαντικά η κάθε οικονομία, παρόλο που έληξε η κρίση, εξακολουθούν να παραμένει η ανάπτυξη χαμηλή σε κάποια κράτη-μέλη και, και κάποια κράτη-μέλη θέλουν να ζήσουν πέρα από τα έσοδά του. Ε, και θα πρέπει να ακολουθηθεί σωστή προσέγγιση για αύξηση της ανάπτυξης. Ο σκιώδης ηγητής Ρόμπερτς πιστεύει ότι το χαμηλό έλλειμμα και το χρέος, χαμηλό χρέος, καθώς και συνετής δημοσιονομικός σχεδιασμός είναι προϋποθέσεις για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε εδώ σήμερα αυτό το θέμα που συζητούμε τα δημοσιονομικό σύμφωνο, σημαντική συμφωνία για δημοσιονομική πειθαρχία που υπέγραψαν τα κράτη-μέλη μετά την χρηματοπιστωτική κρίση αυστηρότερη εκδοχή του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Η οδηγία του Συμβουλίου που προτείνεται εδώ σήμερα θα ενσωμάτωνε το άρθρο 3 τη συνθήκη για στερότητα, συντονισμό κλπ. στο νομικό πλαίσιο όπω ε, σχολίασε και, ε, σχολίασαν και συνάδελφοι και οδηγητέ. Ε, όσον αφορά την έκθεση του συναδέλφου Χούμπνερ, ο κύριος Ζήλε καλωσορίζει ότι είναι περιεκτική και σύντομη, κάτι πολύ ενδιαφέρον για αυτό το κοινοβούλιο καλά στοχευμένη έκθεση. Όσον αφορά τι τροπολογίε, ο κ. Ζήλε καλωσορίζει την προσπάθεια αποσαφήνιση κάποιων σημείων. Κάποιο συγκεκριμένο θέμα θέλει να αναφέρει. Σημειώνει ότι ο εισηγητή προβάλλει ένα επιχείρημα για τη δημιουργία άλλων ενός θεσμού για συνετή δημοσιονομική διαχείριση μες του κανονισμού, παρόλο που ο κανονισμός 473 ε, προβλέπει κάτι τέτοιο ήδη. Διαφωνεί και ο Ζήλε με την ερμηνεία του συγητού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή τη. όχι μόνο δεν δίνει εντολή για τη δημιουργία άλλου, ενό, θεσμού, αλλά αντιθέτω μάλιστα. Σημειώνει και παραθέτω ότι η οδηγία είναι απίθανο να απαιτήσει νέε δομέ και μετά βλέπουμε ότι εδώ μια νέα δομή δημιουργείται. Όμως μια ανακατάταξη των θεσμών των υφισταμένων ίσα χρειάζεται σε κάποια κράτη-μέλη αυτή είναι και η άποψη του κυρίου Ζήλε. Γι' αυτό το σκοπό φρονεί ότι συγκεκριμένες τροπολογίες θα μπορούσαν να διευκρινίσουν τη διατύπωση. Άλλες βελτιώσεις όσον αφορά το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη σύσταση ε, ενό δημοσιονομικού συμφώνου ίσως είναι κάτι απαραίτητο και προσβλέπει ο κύριος Ζήλε σε μια επικοδομητική συνεργασία με τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω μιλητές από την Άλτε. Πάμε στους πρασίνους. Ο Φίλιπ Λάμπερτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποθέτω ότι οι φιλελεύθεροι σε ένα πνεύμα εξοικονόμηση ενεργεία θεώρησαν ότι καλύτερο να ήταν να μην έχουν συζητήσουν για ένα χαρτοφυλάκιο για το οποίο δεν θέλουν να τοποθετηθούν. Αυτό το καταδικάζω, μάλλον το καταδικάζω. Θεωρώ ότι δείχνει δημοκρατικό έλλειμμα. Ε, είναι σημαντική αυτή η νομοθεσία που πρέπει να ευθυνθεί αποκλειστικά από το Συμβούλιο. Δεν αρνούμε στο Συμβούλιο την νομιμότητα, πόρα απέχει άποψή μου από αυτή, αλλά γνωρίζουν πολύ καλά ότι καμιά φορά είναι πιο εύκολο να αναλαμβάνονται αποφάσει που πάνε αντίθετα προ το κοινό συμφέρον με κυκλισμό των θυρών, πατά ανοιχτά, όπω συζητάμε εμεί. Συμφωνώ μαζί σου, Σάντορ. Ε, χρειάζονται υγιή δημοσιονομικά. Αλλά αν θέλουμε υγιή δημοσιονομικά, χρειάζονται και υγιή ε, ιδιωτικά οικονομικά. Και αν κάνουν τι που κάνουν στον ιδιωτικό τομέα, ε, οδηγούμεθα στη χρηματοπιστωτική κρίση και μετά ιδιωτικό τομέα ζητά από το δημόσιο τομέα ε, να του σώσει. Δεν πρέπει να εκπληκθούμεθα ότι μετά από αυτό υπάρχουν προβλήματα δημοσιονομικά. Το μόνο παράδειγμα, το μόνο παράδειγμα από τα δημοσιονομικά ε, είναι η Ελλάδα. όπου, όπου φταίει αυτό. Σ' άλλα ήταν οι υπερβολή του ιδιωτικού τομέα σε άλλε χώρε. Η μόνη εξαίρεση ήταν η Ελλάδα. εκεί η υπερβολική χρέωση του ιδιωτικού τομέα δημιούργησε την κρίση. Αν θέλουμε δημοσιονομικούς κανόνες οι οποίοι να είναι εφαρμόσιμοι θα πρέπει οι κανόνες να είναι λογικοί και να στηρίζονται συνεπώ επί των οικονομικών επιστημών, όχι επί τη θρησκεία, αν θέλετε, τη οικονομική, επί τη επιστήμης. Η επιστήμη όμω, ακυρώνοντας αυτό που μα λένε ότι πέρα από το 60% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέο είναι μη βιώσιμο. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε και περίπτωση της Ιαπωνίας. 200% του ΑΕΠ τη στιγμή που ε, ε, έχουν οι τοπικοί φορείς την ιδιοκτησία αυτή ε, και, χρηματοδοτούν τις κοινωνικά ωφέλιμες επενδύσεις τους. Θα πρέπει να έχει νόημα λογικό κανόνα στο 3% και το 60% ήταν επιλογές απόλυτα πολιτικού χαρακτήρα που δεν έχουν καμία επιστημονική βάση, καμία. Δεν υπάρχει δράμη ε, επιστημονικής προσέγγιση αυτά. Να μην μα κάνουν να πιστεύουμε ότι το 3 και το 60% είναι εξίσου σοβαρά στοιχεία όπω η, έκθεση η χθεσινή που μα έλεγε ότι πηγαίνουμε προ 2 ή 3 βαθμού, 4 βαθμού αύξηση θερμοκρασία στο, στον, ε, στον πλανήτη. Αυτοί έχουν την επιστήμη στο πλευρό του, οι οικονομολόγοι όχι σε αυτή την περίπτωση. Είναι αρκετά παράδοξο που βλέπουμε ότι ενισχύσαμε τους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης στη στιγμή όπου ο το έλλειμμα το δημοσιονομικό συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, από 3,7% του ΑΕΠ πήγε στο 0,9% σήμερα, με τους παρόντες κανόνες, όχι με νέους κανόνες. Δηλαδή μας λένε ότι οι κανόνες δεν λειτουργούν, αλλά βλέπουμε ότι μείωσαν το έλλειμμα. Οπότε είμαστε πολύ πιο κάτω από το όριο του 3%. Και όπω είπε πολύ καλά η Περβάμ Περές, ε, ε, υπάρχουν αυτοί που πλήρωσαν όμω το τίμημα τη πολιτική. Μετά το διαπιστώνουμε και λένε, λέμε δεν υπάρχουν πλέον δημόσιε επενδύσει, λέμε «Ναι, Τι θέλετε λοιπόν, αν κάνουμε αδύνατε τι δημόσιε επενδύσει, αν έχουμε κανόνε λογιστικού που καθιστούν αδύνατε τι δημόσιε επενδύσει, αντίθετα, ε, ε, πολύ καλά γίνεται συνεργασία δημόσιου ιδιωτικού τομέα όπω στην Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί εκπλησόμεθα. Από τη στιγμή που όχι μόνο υπάρχει κατακαιρματισμό κοινωνικό που εμβαθύνεται καθημερινά στην Ευρώπη, αλλά μας λένε ότι θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις 3 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή εκατομμύρια δισεκατομμυρίων ευρώ, για να ανταποκριθούμε στην προκλήση του κλίματος. Όταν τους που λένε ότι περιμένετε μπορούμε να κάνουμε εκείνο παρά μόνο αν πάει καλά η οικονομία. Εγώ θα σας έλεγα, ακούστε παιδιά, όταν δεν υπάρχουν πλέον ανθρώπινα όντα, μην ανησυχείτε, θα υπάρχει πλέον και οικονομία. Λοιπόν, δεν έχει νόημα να λέμε θέλουμε να σώσουμε την οικονομία, σκοτώνοντα τι ίδιε συνθήκε ύπαρξη των κοινωνιών μα στον πλανήτη. Άρα είναι προφανέ ότι χρειαζόμαστε κανόνε δημοσιονομικού. Είναι σαφέ όπω χρειάζονται κανόνε που διέπουν και το, το ιδιωτικό χρέο. Διαφορετικά, αν αφήσετε τα ανθρώπινα όντα να, να μπορούν να φερούν τα πάντα από τη, από τη φύση, θα το κάνουν και από την κοινωνία. Χρειάζονται κανόνε όμω. Οι κανόνε διακυβέρνηση οικονομική Ευρωπαϊκή έχουν σήμερα απεδείχθησαν ε, απέδειξαν ότι δεν είναι σε θέση, είναι σε θέση αδυναμίας να τακτοποιήσουν τις οικονομίες μας, την κοινότητά μας και το περιβάλλον και να θέσουν όλα αυτά ε, σε σωστό μονοπάτι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξαντάσουμε το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι η πρόταση που έχει υποβληθεί δεν κάνει τίποτα, τίποτα, τίποτα για να πετύχει το στόχο. Και θα έλεγα και το εξή. Καμιά φορά διαβάζω το κείμενο και μα τρελαθήκαν αυτοί. Ε, τρελάθηκαν τελείω. Είδαν χτε το Σαλβίνι και τη Λαπέν να πηγαίνουν κατά των οχυρών των Βρυξελών. Και εδώ θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτόματους μηχανισμούς που αρχικυκλώνουν εντελώς τα εθνικά κοινοβούλια, που είναι αντιπροσωπούν τους λαούς, για να λάβουν αποφάσεις, οι οποίες πρώτα απ' όλα είναι αποφάσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα, προϋπολογισμού. Ο βασιλιάς που βασίλευε δια, με απόλυτη εξουσία ε, ε έπρεπε να ανεχθεί το κοινοβούλιο για να ψηφίσει τους προπολογισμού και τους φόρους δεν γινόταν φορολόγηση χωρίς εκπροσώπηση. Και εδώ, στην νομοθεσία, λέμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα υπερκεράζοντας τα κοινοβούλια για να κατατήσουμε τον προπολογισμό. Καταλαβαίνουμε ότι δίνουμε επιχειρήματα σε εκείνους που θέλουν να επαναλαμβάνουν εσαΐ ότι δεν είναι δημοκρατική Ευρώπη. Θα πρέπει τώρα να τα διορθώσουμε αυτό. Λοιπόν, διαβάζοντα τις τροπολογίες, δεν έχω την εντύπωση ότι ε, τελικά επιτυχάνεται ο σωστός ε, στόχος. Um, Ευχαριστώ. Βλέπω ότι ο κύριος Τόρβαλτς έχει ζητήσει το λόγο. Είστε σκιώδης. Ευχαριστώ, το γνωρίζω ότι είμαι σκιώδης. Μέχρι στιγμής δεν έχω προετοιμαστεί, αλλά θα επανέλθω στον, στον εισηγητή το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ. Η Μαρίζα Ματίας για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φτάσαμε στο σημείο πια που πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για το να συμπεριληφθεί το σύμφωνο ε, το δημοσιονομικό ε, σύμφωνο στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Προέρχομαι από χώρα που πλήρωσε βαρύ τίμημα για τις πολιτικές αυτές η Περβάνς και ο Φιλίπ ε, διατύπωσαν πολλές ανησυχίες, τις οποίες επαναλαμβάνω. Να προσθέσω και εγώ την ανησυχία μου για το δημοκρατικό έλλειμμα της οδηγίας που συζητάμε. Έχει είναι, μείνει ένα απομεινάρι αυτή τη τρέλα που οδήγησε στη λιτότητα σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε για δημοσιονομική πειθαρχία αλλά δεν αφορά ακριβώς αυτό η οδηγία. Νομίζω ότι όλοι είναι υπέρ της, των υπεύθυνων δημοσιονομικών. Αλλά τώρα έχουμε μια, ένα κακό ε, καμουφλάς στις προσπάθειες να παρακαμφθούν οι, αγώνες, οι κανόνες της ε, δημοκρατίας. Επί υπήρχε η δυνατότητα των μη εκλεγμένων οργάνων να κυριαρχούν πάνω στις κυβερνήσεις. Είναι ένα είδος ε, πραξικοπήματος, ε, εξαγωγή πραξικοπήματος σε άλλες ε, χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Αυτές οι ανεξάρτητες αρχές δεν υποτίθεται ότι απλώς επισημαίνουν τις ε, παρεκκλήσεις από τον προπολογισμό. Είχαμε το Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών στην Πορτογαλία, παραδείγματο χάρη. Εδώ μιλάμε για ένα είδος πραξικοπήματος. Επιβάλλονται μέτρα στις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, προωθούνται πολιτικές που δεν έχουν εγκριθεί από το εκλογικό σώμα και οι οποίες κυριαρχούν επί οποιοδήποτε μανιφέστου ή οποιαδήποτε δήλωση στην προεκλογική περίοδο. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει νομιμοποίηση, δεν υπάρχουν και αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών λιτότητας ήταν φοβερά, καταστροφικά. Ε, οδήγησαν σε μείωση της δημοκρατίας. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς ε, προσπαθούμε να το εντάξουμε αυτό στο κοινοτικό δίκαιο. Αυτό το δημοσιονομικό σύμφωνο με τη σφραγίδα της καταστροφής που μόλις σας περιέγραψα. Εξελέγην από μια χώρα η οποία πλήρωσε φοβερό τίμημα στη, λόγω των πολιτικών λιτότητας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ανακάμψει σε κάποιο βαθμό Ε, μετά από τα μέτρα προσαρμογής, τα προγράμματα της Τρόικας. Εμείς αντιστρέψαμε αυτές τις πολιτικές. Οι πολιτικές μας έχουν βέβαια τους περιορισμούς τους ακόμα, αλλά σαφώς είναι πολύ καλύτερες από τις πολιτικές λιτότητας που ίσχυαν προηγουμένως. Καμιά από αυτές δεν αναλύεται στην πρόταση της Κομισιόν, ούτε καν στην έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας. Αυτό το οποίο έχουμε εδώ είναι εντελώς λάθος και επ' αυτού έπρεπε να συζητάμε. Καθώς ε, ο πολιταρχισμός ε, αυξάνει στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα υπονομεύοντας την δημοκρατική κυριαρχία. Αυτό θα επιδίνωνε την κρίση. Μιλάμε για κάτι το εντελώς εκρηκτικό το πακέτο αυτό αντιβαίνει πλήρως την ιδέα της ε, Ένωσης ε, Ισότιμων Εταίρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω προσπαθεί απλώς να πλύνει τα χέρια της, να νύψει τα σχήρα σας. Ευχαριστώ κύριε Ζουβάλη. Ευχαριστώ όσον αφορά την ομάδα μου. Διαπιστώνω ότι το Fiscal Compact από τη φύση του το Δημοσιονομικό Σύμφωνο αποτελεί ένα εργαλείο απαράδεκτο όσον αφορά την δημοκρατική συμπεριφορά και προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Να εισάγουμε τώρα αυτή την νομοθεσία της ευρωπαϊκή Ενώσεως παρά το ότι υπάρχει μια οδηγία που κατά κάποιο τρόπο πετυχαίνει τη μεταφορά το περιεχόμενο της διακυβερνητικής συμφωνίας είναι κάτι που δεν θα διορθώσει και της κρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Κατά την άποψή μου έχουμε προτεραιότητες θεμελιώδεις. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μέσα αντιστάθμισης και επιμερισμού των κινδύνων εντός της Ευρωπαϊκής Ζώνης. Ε, πολύ βασικό αυτό για να λειτουργήσει ε, βέλτιστα αυτός ο χώρος. Ε, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τυφλά τους όρους του Μάστριχ. Το 60%, το 3% όπως είπε και ο Λάμπερτς και το λένε μεγάλοι οικονομολόγοι στον κόσμο και μεγάλοι πολιτικοί της Βόρειας Ευρώπης, Γερμανοί, Αυστριακοί, Ολλανδοί, Φιλανδοί που επιβάλλουν αυτές τις πολιτικές που φέρνουν σε ανταγωνιστικό όφελο στις χώρες τους είναι πολύ επικίνδυνο να επηρεάζονται οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις για κάποιες αποφάσεις που από μία άποψη θα μπορούσαν να προσανατολίζονται ως μεγαλύτερη δαπάνη για να ε, αναπτύξουν λίγο περισσότερο την οικονομία εκεί που υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα, εκεί που υπάρχει οικονομική δυσκολία με λογική στατική που συνδέεται με κανόνες ελάχιστα ευέλικτους όπως είδαμε στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το Six Pack και μετά με το Fiscal Compact. Ένας θα έλεγε ότι προσπαθούν μανιωδώς να μειώσουν ακόμα την έννοια της δημοκρατίας και την επιρροή που μπορεί να έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες έναντι του όλου εγχειρήματο. Αυτή η οδηγία, επαναλαμβάνω, έχει τροποποιηθεί στον αφορά την αρχική των 100 μελών και πρέπει να απορριφθεί και η πρόταση τη εισηγήτης πρέπει να απορριφθεί, να τροποποιηθεί η νομική βάση, μετά στο Συμβούλιο να χρησιμοποιηθεί ειδική πλειοψηφία και όχι ομοφωνία. Αυτό είναι κάτι που κατά τη δική μα άποψη θα οδηγούσε να γίνει αποδεκτό κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει και στο τέλο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα πλαίσιο κοινωνικό όπου οι χώρε του Νότου με την επόμενη κυκλική κρίση που θα συμβεί σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να υποχρεωθούν να βάλουν από μέσα το σύστημα που δεν μπόρεσε να οδηγήσει σε επιμερισμό των κινδύνων πριν ε, ζητήσουν μια μείωση που τυφλώνει. Ε, διότι το βάρος θα βαρύνει πάρα πολύ τις κοινωνίες, ε, τους λαούς, τους ανθρώπους που θα αντιδράσουν βία ψηφίζοντας ίσως και πολιτικές δυνάμεις που κατανόησαν τον όλο μηχανισμό και ζητούν πέρα τη δημιουργία και μηχανισμό πυρισμού των κινδύνων και λύσεις για να διαλύσουν την Νομισματική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα χρειάζεται μεγάλη υπευθυνότητα. Δεν, πρέπει να, δεν θα πρέπει να οδηγηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, διότι θα συγκρουστούν οι ευρωπαϊκοί λαοί, θα τους οδηγήσουν προς τα εκεί. Και αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα στοιχείο που διχάζει και δεν ενώνει ε, αυτό το δημοσιονομικό σύμφωνο, το Fiscal Compact. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο Catch the Eye. Ο Μάρκους, εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα πολύ υπομονετικά τη συζήτηση. Εξεπλάγει. Δεν μιλάμε για αναδιαπραγμάτευση του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Αντίθετα, λέμε, εάν ε, ε, διαρωτόμαστε αν το ε, δημοσιονομικό σύμφωνο θα πρέπει να μείνει ως διακυβερνητική συμφωνία ή να ενταχθεί στο κοινοτικό δίκαιο. Μπορούμε να ξαναρχίσουμε ολόκληρη όλη τη συζήτηση αν θέλετε. Αυτή τη στιγμή όμως οι χώρες που έχουν τεράστιο χρέος προσπαθούν να δημιουργήσουν μεγάλη μετατόπιση, μεταφορά πλούτου και διαρωτώ με αν είναι λογικό, είναι σωστή η κοινωνική πολιτική αυτή. Παίρνεις δηλαδή τα χρήματα από τους φορολογουμένους και τα περνάς σε κάποια άλλη κοινωνική ομάδα με τη μορφή πληρωμών. Είναι κρίμα να υπάρχουν τόσο ψηλά επίπεδα φορολόγησης μόνο και μόνο για την εξυπηρέτηση του χρέους. Πρέπει ε, το οικονομικό μας μοντέλο να μας επιτρέπει να χρηματοδοτήσουμε το κράτος πρόνοιας μας. Δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα έχει θεωρήσει ότι το ευρώ είναι ξένο νόμισμα ή ότι αντιμετωπίζεται ως ε, ξένο νόμισμα. Η εθνική οικονομία δεν επηρεάζει το ευρώ ως νόμισμα. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να κάνει ή να μην κάνει ό,τι επιθυμεί. Ε, επειδή οι αποφάσεις της α χώρας μπορεί να επηρεάσουν τις άλλες. Αυτό αποτελεί ε, περιορισμό της ελευθερίας, διότι πρέπει κανείς να αναλαμβάνει και κάποια ευθύνη. Δεν σκέφτεται μόνο τη χώρα του, αλλά και τους εταίρους σου. Δεν μπορεί να θεωρήσουμε ότι είμαστε στον παλιό καλό καιρό όπου μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τους ε, ε, μοχλούς της οικονομικής πολιτικής όπως θέλαμε. Όχι. Ένα μέρος της κυριαρχίας έχει μεταφερθεί στο νόμισμα Και ίσως αν ε, το σκεφτείτε έτσι, ε, τότε τα πράγματα θα είναι πιο ενδιαφέροντα. Αν όμως απορρίπτεται αυτή την ε, οδηγία, και πιστεύετε ότι ο κόσμος θα γίνει καλύτερος και θα ε, επικρατήσει κοινωνική δικαιοσύνη, πλανάστε, διότι η διακυβερνητική ε, συμφωνία μεταξύ κυρίαρχων κρατών θα συνεχίσει να ισχύει. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσει να είναι διακυβερνητική ε, ή κοινοτικό δίκαιο. Τίποτα παραπάνω δεν είναι αυτό, από αυτό. Προσβλέπω στην επερχόμενη συζήτηση, παρά τα αυτά όμως θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε σε αυτό περί του οποίου πρόκειται και βεβαίως ε, δεν θα υπάρξει καλύτερη ευκαιρία. Αυτά ε, θα ακούσετε από τη θέση που αυτόν αυτών που έκαναν τόσο ηχηρές ομιλίες σήμερα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έχω κι εγώ χρόνο να πάρω το λόγο. Ή μπορεί να ζωηρέψει η συζήτηση. Έχω κι εγώ δικαίωμα να μιλήσω στον χρόνο του Catch the Eye. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, είναι καλό που γίνεται. Είναι και λίγο παράδοξη βέβαια, καθότι η οδηγία δεν ε, ενσωματώνει μόνο το σύμφωνο αυτό ε, στην Ένωση, αλλά εισάγει και κάποιες μικρές και κάποιες αλλαγές. Θα ήθελα λοιπόν να επισέλθω ε, στην ουσία. Έχουμε όμως δύο σημεία τώρα που, για τα οποία, των οποίων υπάρχει αντιπαράθεση. Το ένα είναι προφανές. Δεν μπορεί να έχουμε κοινό νόμισμα αν δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες, μια κοινή βάση. Ε, ε, που να είναι ευέλικτοι αλλά που να μην μπορούν να παραβιάζονται. Αυτό είναι δύσκολο να το αμφισβητήσει κανείς. Η άλλη πλευρά που δύσκολα επίσης και αυτή αμφισβητείται είναι ότι οι κανόνες που έχουμε τώρα είναι τέλειοι, είναι καλοί για κάποια οικονομική πολιτική. Και εγώ πολύ δύσκολα μπορώ να συμφωνήσω με κάτι τέτοιο. Αυτό έχει αποδειχθεί έχει αποδειχθεί πολύ καλά ότι δεν ισχύει και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όταν εισάγεται μεγαλύτερη ευελιξία. Είναι λοιπόν σαφές ότι οι διατάξεις ως έχουν ε, είναι υπερβολικά ε, κυκλικοί και δεν αντιμετωπίζουν ε, τις δυσκολίες, την περίοδο των δυσκολιών. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο ως αφετηρία. Κάτι που είπε ο Μάρκος ισχύει. Πρώτον, ό,τι και να κάνουμε με την οδηγία, και όχι μόνο, όχι μόνο το δημοσιονομικό σύμφωνο υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά θα εξακολουθήσει να υπάρχει και το σύμφωνο σταθερότητας, γιατί το σύμφωνο ε, το δημοσιονομικό σύμφωνο δεν ζητά μόνο να ε, εισάγουν τα κράτη-μέλη και της νομοθεσία αλλά και το ε, σύμφωνο σταθερότητας de facto θεωρείται ότι ο ισοσκελισμένο προπολογισμό είναι αυτός που τον ερμηνεύει ω τέτοιο η Κομισιόν. Αν ε, ισχύσει τώρα η ευελιξία, αυτό ισχύει και στο πλαίσιο του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Έχουμε λοιπόν το SGP και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Τι ε, γίνεται με αυτό είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν αρκεί και έχει πάρα πολλά προβλήματα για να το πάρουμε ως έχει. Η πρόταση τροποποιεί και αλλάζει όλο το άρθρο 3, εγώ έτσι το ερμηνεύω φυσικά, δεν μπορώ να συζητήσω καν αν δεν ε, ξεκαθαριστεί αυτό, και είναι σαφές ήδη από τις ε, αιτιολογικές, ε, από τα ε, εκτιμώντας. Και κάπου στο άρθρο 3.1α αναφέρεται ένας ε, μικρο, με, μεσοπρόθεσμος στόχος. Δηλαδή αυτή η πρόταση δεν είναι καταρχήν ασυμβαστή με έναν άλλο μεσοπρόθεσμο στόχο το 0,1 του Συμφώνου Σταθερότητας και μετά έχει ε, εισαχθεί το 0,5 για τις ε, χώρες με μεγάλο χρέος. Αλλά ποιο είναι το νόημα. Η οδηγία το κάνει αυτό σε αντάλλαγμα περισσότερο δεσμευτικών μεσοπρόθεσμων κανόνων επί του χρέους, που και αυτό μπορεί να είναι ένα αντιστάθμισμα. Σου προσφέρω ευελιξία για να καθορίσεις τους ε, καθορισμένους ε, στόχους σου μεσοπρόθεσμα, αλλά άπαξ και δηρείς αυτό το δρόμο πρέπει να τον τηρείς. Αυτό, αυτή η αντισταθμιστική προσφορά μπορεί να έχει νόημα καταρχήν, όχι όπως έχει διατυπωθεί, αλλά ενδεχομένως να το ελάβαινα υπόψη μου. Αλλά η ουσία ποια είναι, ότι αν δεν τροποποιηθεί εκ παραλίλου το σύμφωνο σταθερότητα και αν δεν δώσεις νόημα σε αυτό που λέει εδώ ένας μεσοπρόθεσμος στόχος και πει ο μεσοπρόθεσμος στόχος συνεπάγεται σκελισμένο προπολογισμό, τότε αυτό μένει κενό γράμμα. Δεν υπάρχει αλλαγή και υπάρχει μόνο η επιπλέον αυστηρότητα σχετικά με τη συμμόρφωση του Μεσοπρόθεσμου Συμφώνου και της ε, δημοσιονομικής αυτής αρχής που μπορεί να παρέμβει στην δημοκρατική διαδικασία που είναι λίγο ωριακή όσον αφορά τα συντάγματα. Για να υπάρχει αντιστάθμισμα που να έχει νόημα σημαίνει ότι κάτι σου δίνω και παίρνω κάτι σε αντάλλαγμα. Αντί λοιπόν και αν δεν αλλάξει λοιπόν το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης δεν θα έχουμε ε, ανταλλάγματα. Αν δεν ε, εκ παραλίλου ανοίξει το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης δεν θα γίνει αποδεκτό. γιατί θα συνεχίσουν να ισχύουν και τα δύο σύμφωνα ως έχουν αν δεν γίνει καμιά αλλαγή. Αυτό που είπε ο Μάρκος ισχύει απολύτως. Με την απόρριψη δεν αλλάζουμε τίποτα επί τα βελτίο. Όμως ισχύει ότι αν δεν υπάρχει κάποια συναλλαγή τότε θα έχουμε ε, ε, ε, μια επιπλέον αυστηρότητα χωρίς το αντάλλαγμα για να είμαι δίκαιος απέναντι στην Επιτροπή υπάρχει. Αυτό είναι καλύτερο ε, κείμενο από ότι το αντίστοιχο άρθρο του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Προσωπικά λοιπόν θεωρώ ότι χωρίς τροποποίηση, χωρίς αναμόρφωση του Συμφώνου ε, αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό για να συνεχίσουμε. Και αυτό δεν θα αλλάξει τη νομική βάση, γιατί αυτό ήταν ένα πολύ έξυπνη τρόπος, ε, καταλαβαίνω, η Ντανούτα να ξεπεράσει την, ε, το εμπόδιο της ομοφωνία, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Αυτό το άρθρο, αυτή η οδηγία υποκαθιστά το άρθρο 3 του, συμφώνου, του Δημοσιονομικού Συμφώνου, το οποίο είχε ε, γίνει σε διακυβερνητική διαδικασία. Γιατί, Γιατί ο Κάμερον είχε αντίρρηση με την προτινόμενη τροποποίηση του ε, και τότε ο, ο ε, Ρομπαϊ ε, είχε προτείνει να γίνει στην παράγραφο 2 και όχι στην 3. Το να γίνει αυτό παράγραφος 3 αποτελεί σημαντική αλλαγή γιατί αλλάζει όλη την ουσία, την αρχική ουσία του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Και από ιστορική άποψη αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ποτέ δεν θα δεχτούμε αυτή τη νομική βάση. Γιατί θα αλλάξει το όλο θέμα από την αρχή. Δεν είναι λοιπόν μια απλώς διαδικαστική τροπολογία. Είναι υποκατάσταση του Δημοσιονομικού Συμφώνου που ευθύς εξ αρχής είχε θεωρηθεί ε, ως ε, σημαντική προσθήκη στο πρωτόκολλο γιατί το πρωτόκολλο δεν αναφέρεται πουθενά η διάταξη για τον ισοσκελισμένο προπολογισμό μόνο το 3 και 6%. Έτσι πρέπει να, ε, να προσθέσουμε μια τρίτη παύλα. Άρα είναι ουσιαστική ε, τροποποίηση του πρωτοκόλου και ω εκ τούτου δεν το δέχομαι για την παράγραφο 3, πρέπει να παραμείνει στην παράγραφο 2. Εξαιρετικά χρήσιμη συζήτηση, καλό είναι που την κάνουμε και αυτή θα πρέπει να γίνει ακούγοντα ο ένα το επιχείρημα του άλλου και όχι απλώ να ε, προβάλλουμε την αλήθεια που θεωρεί ο καθένα μα ότι έχει. Βεβαίω είναι προφανέ και το ίδιο ισχύει και στο Συμβούλιο, όλοι γνωρίζουν ότι το θέμα αυτό δεν θα προχωρήσει προ το παρόν το γνωρίζουμε και ας το χρησιμοποιήσουμε για βάση, για μια συζήτηση, όμως το θέμα αυτό, το οποίο είναι πολύ λεπτό, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μέχρι ότου ολοκληρωθεί με τρόπο ολοκληρωμένο. Η στιγμή δεν είναι κατάλληλη, ο χρόνος δεν έχει οριμάσει και απέναντι στον Μάρκο Βάλλη, ο τρόπος με τον οποίο εσύ και η κυβέρνησή σου, η, προ... η πλειοψηφία σου αντιμετωπίζει το πρόβλημα των δημοσιονομικών κανόνων, βλάπτει οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωση των κανόνων, γιατί τον αμφισβητεί κανείς τους απολύτως λογικούς Κανόνε κανόνες ε, οδηγεί στο να σκληρύνει έτσι περαιτέρω η θέση αυτών οι οποίοι είναι αντίθετοι. Αυτή είναι, αυτός είναι ο χρυσός κανόνας. Πρέπει λοιπόν η συζήτηση να γίνει ευφιέστερη με τρόπο που, ώστε ο καθένας να ακούει τον άλλον. Γιατί πάντοτε σε αυτές στις θέσεις ακόμα και του πιο σκληρού αντιπάλου υπάρχει κάποιος ε, κόκος αλήθειας. Ε, να, να ακούσουμε ε, αν δεν ακούσουμε αυτή τη βασική αρχή, αν δεν την ακολουθήσουμε, δεν θα οδηγηθούμε πουθενά. Αντίπαλος... Ε, ε της ε, Ιταλικής Λέγκα και των Πέντε Αστέρων. Και τώρα ο κύριος Μάννα. Ε, λοιπόν, πολύ παθιασμένη η ομιλία. Συμφωνώ. Ήταν χρήσιμη η συζήτηση, είναι χρήσιμη η συζήτηση. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να εξετάσουμε τις διαφορές οι οποίες είναι απολύτως ε, ουσιαστικές. Ο Μάρκος Βέμπερ έχει δίκιο. Δεν αμφισβητείται το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Όμως αν δούμε ότι για ποιο λόγο χώρες όπως η Γερμανία όπου υπάρχει μια απολύτως ε, σόφρον πολιτική αποταμιεύσεων, όπου έχει υπάρξει απαγόρευση στον προπολογισμό, που ήταν απολύτως λογικός, λογική αυτή η απαγόρευση, σημαίνει ότι μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε χρήματα και να τα επενδύσουμε. Αυτό είναι θετικό για τον κόσμο. Επίσης, βεβαίως, το Σύμφωνο Σταθερότητας πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο. Αλλά με αυτούς που λένε ότι πρέπει να το καταργήσουμε δεν συμφωνώ. Γιατί υπάρχουν κάποια κράτη όπου λειτουργεί η οικονομία και αυτό δεν είναι τυχαίο. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε κάποιους μηχανισμούς για να επιτύχουμε και λογικά αποτελέσματα. Ας ε, κάνουμε ένα βήμα πίσω, πίσω για να μην κάνουμε λάθος εκτιμήσεις. Και είναι σωστό επίσης ότι οι διακυβερνητικές, οι διακυβερνητικές λύσεις δεν ε, λειτουργούν γιατί πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις με ε, ομοφωνία και πρέπει να περάσουν όλα αυτά στην κοινοτική μέθοδο. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή χαιρετίζεται στην Ιταλία ε, είναι εντελώς λανθασμένο. Να λέτε ότι τότε αποφασίζεται στην, ε, ε, στις Βρυξέλλες το αγνοούμε, κάνουμε υποσχέσεις που δεν πρόκειται να τηρηθούν και δεν μπορούν να τηρηθούν. Αλλά στην ουσία Θεωρώ ότι αυτός είναι ο πιο λανθασμένος τρόπος. Και υπάρχει και ένα σαφές μήνυμα. Όταν ε, μπαίνει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κράτη-μέλη εγκαταλείπουν ένα τμήμα της κυριαρχίας του και μάλιστα εθελουσίως. Γιατί θέλουν να ενταχθούν στην Ένωση. Ορισμένες παρατηρήσεις που γίνονται ε, πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη στο γενικότερο πλαίσιο. Το ευρώ είναι ένα εγχείρημα για να υπάρξει ειρήνη. Εντάξει. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κάνουν ε, διάφορες χειρές ε, δηλώσεις για να πάρουν κάποιο χειροκρότημα όταν συζητούν με τους φίλους τους. Βεβαίω πρέπει να γίνονται και αυτές οι συζητήσεις, αλλά το βασικό είναι να συνεχιστεί η σοβαρή συζήτηση. Και δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε αυτά που επιτύχαμε. Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα και δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα μιμηθούμε όλα. Αλλά πρέπει να ερωτηθούμε γιατί ορισμένα πράγματα πάνε καλά. Γιατί ελέγχεται ο προπολογισμό, γιατί τότε μπορούμε να επενδύσουμε και τότε μπορούμε ακριβώ να ε, χρηματοδοτήσουμε και τα απαραίτητα κοινωνικά μέτρα. Αυτή είναι μια πολύ λογική κοινωνική οικονομία της αγοράς. Ευχαριστώ, λέει Και τελευταία η Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω επεμβαίνω ξανά στη συζήτηση, θεωρώ ότι δεν είναι καλά τοποθετημένη. Εδώ δεν μιλάμε για το Μισονικό Σύμφωνο, δεν κάτι μικρό. Πρέπει να θυμηθούμε πώς υιοθετήθηκε. Και ας θυμηθούμε, θέλαμε να έχουμε σωστή προσέγγιση. Διαφορετικά, δεν θα το είχαμε. Έχουμε νομικό πλαίσιο που καθορίζεται με το 6-pack και το 2-pack. Βάσει αυτού λειτουργούμε. Να θεωρούμε σήμερα ότι μπορούμε να ανοίξουμε και έχω υπόψη μου το ρόλο του Κοινοβουλίου. Θέλουμε τουλάχιστον αυτό το σύμφωνο να πάψει να είναι ένα εργαλείο απλώς διακυβερνητικό. Να μπορεί να ενταχθεί στο κοινοτικό πλαίσιο. Αλλά λέγαμε πάντα στους σοσιαλιστές ότι για μας αυτή η ένταξη, αυτή η ολοκλήρωση δεν μπορεί να γίνει χωρίς αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος. Βέβαια, το επανελέμβανα και όταν συζητούσαμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ο καθένας πρέπει να σέβεται ένα κώδικα, οδικό χάρτη, τους κανόνες για τη συνδιοκτησία του ευρώ. Αλλιώς δεν θα αντέξει το ευρώ. Αυτή είναι η βάση του ενίου νομίσματος αλλά έχουμε κάποια δεδομένη στιγμή το δικαίωμα να δηλωτηθούμε όσον αφορά τη σκοπιμότητα της λειτουργίας των κανόνων. Κατανοώ αυτό που είπε ο Τόμας Μαν. για το μηδενικό έλλειμμα. Και διερωτώ με, τι αντίκτυπο είχε στην ευρωπαϊκή οικονομία αυτό. Αυτή η Επιτροπή ξεκίνησε με το σχέδιο Juncker. Τι είναι το σχέδιο Juncker. Γιατί το είχαμε, όχι για να τον ικανοποιήσουμε τον κύριο Γιούνκερ, διότι οι κανόνες οικονομικής διακυβέρνηση δεν απαγορεύουν σε μια οικονομία τόσο σημαντική όπως είναι η Ευρωζώνη να έχει ένα επίπεδο επενδύσεων που θα προσαρμόζεται λίγο πολύ στις ανάγκες της Ευρωζώνης και θα επιτρέψει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της. Δεν θέλω να ξεχωρίσω τη Γερμανία. Κάθε φορά όμως που πηγαίνω στη Γερμανία διαπιστώνω ότι το θέμα των δημοσίων επενδύσεων είναι επιτάπητος. Και όλοι το συζητάνε. Δεν είναι ότι επειδή είναι μια χώρα σε πλεόνασμα που δεν θα τεθεί αυτό το ζήτημα. Ο στόχος μιας οικονομίας δεν είναι αποκλειστικά να έχει πλεόνασμα και να πουλά αυτοκίνητα στη Γερμανία. Να εξασφαλίζει και την, ε, το, στο ε, κατάλληλο επίπεδο διαβίωση για όλους τους συμπολίτε είναι ένας από τους στόχους οικονομίας. Συ... Συγγνώμη που τη Γαλλία. Δεν είναι καλό μιλάει ένα Γάλλο για τη Γερμανία, ούτε το αντίστροφο είναι πάντα καλό. Εκτό όταν συμφωνούμε. Πριν συμφωνήσουμε όμω, θα πρέπει να θέσουμε επιτάπητο στα προβλήματα. Αναγνωρίζω ότι η χώρα μου δεν είναι πάντα υπόδειγμα όσον αφορά τη μείωση του δημοσίου ελλείμματος, όσον αφορά τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών. Από την άποψη όμω τη βιωσιμότητα των δημοσίων επενδύσεων, νομίζω ότι τίθεται το θέμα. Σε αυτή τη θητεία δεν μπορούμε απλώς σαν διοικητική πράξη να εντάξουμε αυτό το σύμφωνο εντός του κοινοτικού δικαίου χωρίς να δούμε κατά πόσο είναι σκόπιμοι οι κανόνες οικονομικοί και πολιτικοί που ακολουθούμε. Επ' αυτού η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπολείπεται του απαιτουμένου. Και θα πρέπει να διορθώσουμε τις προπτικές που προτείνει η εισηγήτρια. Διότι αν το κάνουμε αυτό θα χάσουμε την ευκαιρία. Δεν θα μπορούμε να είμαστε ε, δίκαιοι, σωστοί από πλευράς νομικής εάν προσεγγίσουμε το ζήτημα με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής. Εκτός αν θέλετε να μιλήσετε. Αν θέλετε. Όχι. Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξή. Προθεσμία για τι τροπολογίε 18 Οκτωβρίου, συζήτηση τροπολογιών 12 Νοεμβρίου. Ψηφοφορία στην Οίκον. Έτσι προγραμματίζει η συγγήτρια τουλάχιστον. Υπάρχουν δισταγμοί γι' αυτό, θα δούμε. 27 Νοεμβρίου του 2018. Επόμενο θέμα. Ετήσια έκθεση για την Τραπεζική Ένωση. Τόμας Μάν είναι ο εισηγητής. Όχι. Τόρβαλς. Νίλ Τόρβαλς. Σκιώδης εισηγητής. Είναι ο Τόμας Μάν. Συγγνώμη Νίλ. Έχεις το λόγο Νίλ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι και ο Τόμας δεν ήταν ε, εξαίρετος εισηγητής. να δούμε το παρελθόν. Γιατί συζητήσαμε και για αυτό το δημοσιονομικό σύμφωνο που και αυτό ε, ασχολήθηκε με το παρελθόν. Στο τέλος δεκαετίας του 60 θα θυμάστε κατά τη συνάντηση κορυφής στην Χάγη ο Βίλι Μπραντ είχε μια καινούργια ιδέα. Οι Γερμανοί επειδή είχαν εμποχτήσει να τους πιέζουν πάντα με τον ίδιο τρόπο, επειδή είχαν μαζί με τους Ολλανδούς πιο δυναμική οικονομία, κάθε τόσο ανατιμούσαν το νόμισμά τους και άλλοι έπρεπε να το υποτιμήσουν. Και η κατάσταση αυτή επαναλαμβανόταν. Οπότε ο Βίλι Μπραντ είχε μια ιδέα. Είπε να δημιουργήσουμε ε, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. όπου οι Γερμανοί θα τοποθετούσαν 20% του αποθεματικού συναλλάγματός τους, αλλά με μία προϋπόθεση. Ότι όλοι θα προσπαθήσουν να υιοθετήσουν παράλληλη δημοσιονομική πολιτική. Διότι αν δεν υπήρχε νομισματική και δημοσιονομική πολιτική προς την ίδια κατεύθυνση δεν θα λειτουργούσε. Αλλά ακόμη περιμένουμε ότι χρειαζόμαστε, να καταλάβουν όλοι, ότι χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό Μεσματικό Ταμείο και για να γίνει αυτό όλοι πρέπει να τηρούν τους ίδιους κανόνες γιατί αλλιώς ορισμένοι δεν θα πληρώνουν το εισιτήριό τους και με τσαμπατζίδες δεν γίνεται τίποτα. Ελπίζω λοιπόν σε μερικά χρόνια να γίνει μια λογική συζήτηση για το πλαίσιο. Η Τραπεζική Ένωση είναι πολύ ενδιαφέρουσα αν τη δούμε στο ιστορικό πλαίσιο. Διάφοροι το επέκριναν ε, ιδιαίτερα. Τώρα όμως έχει αποδείξει ότι είναι χρήσιμη. Ας πούμε τι έγινε στη Φιλανδία την προηγούμενη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα. Η μεγαλύτερη τράπεζα της, ε, των χωρών του Βορρά πήγε στο Ελσίνκι, η Νορντέα γιατί λόγω της Τραπεζικής Ενώσης είχαν ένα καλύτερο πλαίσιο από τη Σουηδία. Παρόλο που η Σουηδία θεωρείται ιδιαίτερα σταθερή. Στο σχέδιο εκθεσής μου λοιπόν στέλνω ένα αρκετά θετικό μήνυμα. Όμως δεν έχει πλήρως ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση, να μην το ξεχνάμε. ούτως ώστε από μόνη της να διευκολύνει την ε, σταθερότητα και την ανάπτυξη. Και για να βελτιωθεί η κατάσταση πρέπει να έχει και λογικούς και συνεκτικούς κανόνες ε, και να συνεργάζεται με τις αρχές εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης. Η έκθεση ακολουθεί το παράρτημα, το πρότυπο και των προηγούμενων. Ε, επίβλεψη, εξυγίανση και εγγύηση των καταθέσεων. Και βεβαίω περισσότερο μα ενδιαφέρει να προωθηθούν οι κανόνε κατά του ξεπλήματο χρήματο. Είχαμε πρόσφατα μια υπόθεση στην ε, Φινλανδία. Η αστυνομία έκανε μια επιδρομή σε ένα νησί στη Φιλανδία, σε μια εταιρεία και πίσω από αυτό το τον οργανισμό που στην ουσία εξέπαιρνε χρήμα, βρήκαμε ένα χρυσό, πανε, ε, συγγνώμη, χρυσό διαβατήριο, όπως λέγεται, της Μάλτας. Πρέπει λοιπόν να ε, ξαναδούμε και την ε, προσέγγιση μας για την ε, νομισματική πολιτική. Και η κύρια ευθύνη την έχουν τα κράτη-μέλη και οι ίδιες τράπεζες. Δεν υπάρχει καμία πανάκια που να μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Και αν θέλετε να ξέρετε πώς μπορεί να λυθεί κάθε πρόβλημα, τότε ζείτε σε έναν φανταστικό κόσμο. Πρέπει οπωσδήποτε να προπαρασκευαστούμε για τις μεγάλες αλλαγές, αλλά όσο και να προπαρασκευαστούμε, εμείς δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε την προπαρασκευή που πρέπει να κάνει και ο, και ο ιδιωτικός τομέας. Επίσης, Υπενθυμίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ένα ρόλο επίβλεψης. Είχαμε κάνει μια συζήτηση και με τον κύριο Ντράγκη που είπε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό το ρόλο αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Είναι καλό να παίζει αυτό το ρόλο η ΕΠΣΟΚΑΠΑΤΑΒ για την εξυγίαση. Συμφωνώ ο ESM να γίνει ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και βλέποντας και το ιστορικό νομίζω ότι είναι σκόπιμη, θα ήταν σκόπιμη μια τέτοια εξέλιξη. Αλλά να βασιστεί σε σαφείς προϋποθέσεις για να υπάρχει υπευθυνότητα και να μην υπάρχει ηθικός κίνδυνος. Επίσης τονίζω τους κανόνες της ε, προληπτικής κεφαλαιοποίησης. Αυτά πρέπει να διευκρινιστούν. Επίση, να μην ξεχνάμε την ανάγκη στενής συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤΑΦ και του ενιαίου μηχανισμού εξυγένση και χαιρετίζω τα τελευταία βήματα. Τώρα για το ε, σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Δεν θέλω να παρέμβω στη δουλειά των συναδέλφων που είναι σε διαπραγματεύσεις για αυτό το θέμα, αλλά τονίζω ότι χρειαζόμαστε το έντις ως τρίτο πυλώνα της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Και πρέπει πρώτα να μειώνονται οι κίνδυνοι και κατόπιν να υπάρχει καταμερισμός τους. Δεν πρέπει να αυξάνονται οι κίνδυνοι και μετά να προσπαθούμε να τους μοιράσουμε. Κατά λίγο. Η έκθεση στέλνει ένα θετικό μήνυμα για την Τραπεζική Ένωση και για τα θεσμικά όργανα που πρέπει να την εφαρμόσουν. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ρωμαλαίο σύστημα που θα ενισχύσει την οικονομική μας ανθεκτικότητα και θα μας βοηθήσει να έχουμε περισσότερη ανάπτυξη. Και προσβλέπω στην συμβολή των ε, σκιωδών και των άλλων συναδέλφων. Θα κάνω ό,τι μπορώ και να λάβω υπόψη τα σχόλιά σας και είμαι πεπισμένος ότι θα καταλήξω σε ένα κείμενο που να τύχει στήριξη από την ευρεία πλειοψηφία της Επιτροπής μας και ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ ε, τον εισηγητή. Δίνουμε το λόγο στον Τόμας Μαν, τον πρώτο σκιώδη ηγητή. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι ένας από τους ε, αυτόματους κανόνες ε, που υπάρχουν είναι ότι στις Βρυξέλλες πέφτουν τα, ε, κλείνουν τα παντζούρια γιατί δεν πρέπει να μας βλέπει ο ήλιος. Εν πάση περιπτώσει, αν μπορούσαμε να ανάψουμε κανένα φως. Τόμας Μάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Αυτό, το σκότος όμως δεν ε, συνδυάζεται με την έκθεση. Γιατί η έκθεση είναι πολύ καλή και τον συγχαίρω. Γιατί τα μηνύματα που στέλνουμε είναι σημαντικά. Δεν είναι μόνο θετικά, αλλά είναι και επικοδομητικά, επικριτικά. Θέλουμε η οικονομία μας να αντέχει. Η Τραπεζική Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί λοιπόν. Αυτό είναι ένα βασικό βήμα για μια λειτουργική ενιαία αγορά, για ισότιμο ανταγωνισμό και περισσότερη προβλεψιμότητα για όσους συμμετέχουν στην οικονομία. Όμως δεν θα πρέπει να αυξηθεί ιδιαίτερα το κόστος για τις τράπεζες. Γιατί αυτό θα είχε αρνητικέ επιπτώσει για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και τη χρηματοδότησή του. Πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί η αρχή τη αναλογικότητα. Η Τραπεζική Ένωση πρέπει να γίνει πιο σταθερή βεβαίω. Η εισαγωγή του ΕΝΤΙΣ πρέπει να συνεχιστούν. Σε πολλά σημεία συμφωνώ με τον εισηγητή. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ολοκληρωθεί και η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών Πρέπει να διατηρηθούν ε, τα διαφορετικά μοντέλα για τη λειτουργία των τραπεζών. Αυτό είναι αναγκαίο για τη λειτουργία των οικονομιών μα. Χρειαζόμαστε και συγκεκριμένε διατάξει για το ξέπλυμα χρήματο. Πολλά έχει υποβάλει το Κοινοβούλιο και μέσω των ειδικών επιτροπών και πρέπει να μπορέσουμε να τα επιβάλλουμε αυτά μέσω τη Τραπεζική Ένωση και όχι να αναβάλλονται όλα αυτά όπω μέχρι τώρα. Τα κράτη-μέλη και οι αρχέ επίβλεψη πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούν και με το θέμα των κόκκινων δανείων. Είναι πολύ σημαντικότερο από ό,τι θεωρούσαμε μέχρι στιγμή. Και τέλο, θεωρώ ότι οι αρχέ επίβλεψη πρέπει να ασχοληθούν και με την κύβερνο ασφάλεια. Πολύ σημαντικό θέμα. Το Brexit, ε, ναι, μπορεί να έχει ε, σημαντικές επιπτώσεις, αλλά ε, το βασικό θέμα είναι η ισορροπία δυνάμεων μεταξύ τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ όλων των άλλων κρατών, όλοι οι εμπλεκόμενοι και πάνω απ' όλα οι αρχές επίβλεψης πρέπει να είναι διατεθειμένοι να αντιδράσουν σε διαφορετικά σενάρια, όχι μόνο σε ένα πλάνο Α και πλάνο Β. Και τα κράτη-μέλη που δεν είναι στην Ένωση, την ε, ε, ΟΝΕ, πρέπει να ενθαρρυνθούν να ε, ενταχθούν. Και να και ο ήλιος. Να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να εκλεπτύνουμε τις κεφαλιακές απαιτήσει και τα, οι υπάρχοντες κίνδυνοι πρέπει να ληφθούν υπόψη όσο γίνεται. Αγαπητέ Νίλς, είναι τόσο καλή η έκθεσή σου, αλλά θα κάνω κάποιες προτάσεις για να την ενισχύσω και όχι για την αποδυναμώσω. Νομίζω ότι θα συνεργαστούν πολύ καλά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο Χώνας Φερνάντες από την ομάδα S&D. Ε... Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Α, α, πολύ ευχάριστο που έχουμε ήλιο. Ευχαριστώ τον συγκητή για την εργασία του. Το κείμενο που συζητάμε σήμερα είναι ένα κείμενο που προσανατολίζει καλά τη συζήτηση, είναι λογικό, θα μας βοηθήσει. Φυσικά δεν ε, συμμερίζομαι όλες τις ιδέες που περιέχει, αλλά είναι χρήσιμο για να διαρθρώσει τη συζήτησή μας, για να είναι επικοδομητική και για να καταλήξουμε τους επόμενους μήνες σε συμφωνία. Ποιος είναι ο τελικός στόχος του κειμένου. Είναι να προωθήσει την ολοκλήρωση της, Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Και βεβαίως όλοι αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι ολοκληρωμένη η Τραπεζική Ένωση. Όπως ξέρετε, υπάρχουν ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και έλεγχος όλων των ε, τραπεζικών ιδρυμάτων. Υπάρχει μια εποπτική αρχή όλων των ε, ε, τραπεζικών ιδρυμάτων. Υπάρχει μια αρχή εξυγένσης και ένα ταμείο που επιτρέπει να λαμβάνουν χώρα αυτές οι εξυγιάνσεις. Αν υπάρξει ένα πρόβλημα με μια συγκεκριμένη τράπεζα στο μέλλον, λογικό είναι πέρα από την πρώτη ευθύνη που είναι των ίδιων των διαχειριστών της, πρέπει να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή ευθύνη. Δηλαδή, οι υποπτικές αρχές και οι ρυθμιστικές αρχές γίνονται από ευρωπαϊκές αρχές. Ωστόσο, εάν υπάρξει μια τραπεζική κρίση, όπως είναι τώρα η Τραπεζική Ένωση, τα κράτη-μέλη και οι εθνικές ασφαλιστικές αρχές θα έπρεπε να αναλάβουν σε τελευταία ανάλυση ε, την ευθύνη για να πληρώσουν ε, τις καταθέσεις. Αυτό είναι μια ουσιώδης ανισορροπία. Δηλαδή αυτοί που κάνουν την ε, εποπτεία δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν και τις οικονομικές ευθύνες εάν κάνουν λάθη. Όταν έγινε η πρώτη κρίση μεταξύ του 7 και του 10 οι χώρες οι οποίες έλεγχαν τις τράπεζές τους χρειάστηκαν να αναλάβουν και τις απώλειες. Γιατί η ευθύνη τότε ήταν εθνική της εποπτείας. Τώρα που έχουμε κοινού θεσμού, πολύ δύσκολο θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε στους συμπολίτε μας ότι εσείς πρέπει να πληρώσετε για το ότι οι ευρωπαϊκές αρχές ε, έκαναν επαρκώς τον έλεγχο. Αυτή η έκθεση λοιπόν, σωστά θεωρώ, ε, περιγράφει αυτή την ανισορροπία που υφίσταται στην Τραπεζική Ένωση και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει το κείμενο αυτό να εστιάσει στην αναγκαιότητα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, να υπάρχει μία ίστατη λύση, ένα backstop για την ε, Τραπεζική Ένωση, για να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικέ κρίσεις. Τις επόμενε λοιπόν εβδομάδες που θα συζητήσουμε αυτό το κείμενο, θα υποβάλουμε τις τροπολογίες μας, αλλά τονίζω ότι στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί τάχιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά θα το συζητήσουμε και πιστεύω ότι, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε και ευχαριστώ τον ε, Νίλ Στόρβαλτς και τους υπόλοιπους σκιώδεις που χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συνεργαστώ μαζί τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Ζήλε για το ECR, ο κύριος Λούβετς. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ο Ρόμπερτ ε, ε, ζητά συγγνώμη που λόγω των εθνικών εκλογών στη Λετωνία δεν μπορεί να παρίσταται. Ζητά συγγνώμη ευχαριστεί τον εισηγητή για την προσπάθεια να συνταχθεί μια εξισορροπημένη σε γενικέ γραμμέ έκθεση και κυρίω βρίσκει ε, χρήσιμο το γεγονό ότι η ετήσια έκθεση αναφέρεται στα συγγεγονότα του προηγούμενου έτου, κυρίω όσον αφορά τα θέμα των σκανδάλων για το ξέπλυμα χρήματο και αυτό ε, απαιτεί επιπλέον ε, επιθεώρηση, επίβλεψη. όσον αφορά την ουσία, ο Ρόμπετ πιστεύει ότι η ε, η επίβλεψη τόσο στο τομέα του Prudential όσο και στο AML θα πρέπει να ισχυρθούν και δεν ε, ε, συνάδει με το στόχο της διατήρησης της πολυμορφίας των, μοντέλων, των τραπεζικών μοντέλων της Ευρώπης και τα οποία εκτιμά τη δουλειά που έχει γίνει για την έκθεση αυτή, η οποία είναι ε, ε, σύντομη και ουσιαστική και περιμένει να γίνει συζήτηση. Ο Φίλιπ Λάμπερτς. Ή επί της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Είσαι σκιώδης. Ο, το αφεντικό μου ποτέ δεν μου το είπε αυτό. Ποτέ δεν μου το ανακοίνωσε. Στην ΕΚΟΝ είναι αφεντικό μου. Μια άλλη φορά λοιπόν. Ο Μιγέλ Βιέγα. Εσύ το γνωρίζει, έχει ενημερωθεί. Θα προσπαθήσω να αυτοσχεδιάσω λίγο. Στα πορτογαλικά ο συνήθως. Είναι σαφές νομίζω ότι πρέπει να διατυπώσουμε ανησυχίες. Μας ανησυχεί πολύ αυτή η κατάσταση. Τι βλέπουμε ότι οι βασικές αρχές που υποτίθεται ότι βρίσκονται στη βάση της Τραπεζικής Ένωσης μας δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητά της ε, είναι αμφιλεγόμενη. Πολύ μεγάλες, ε, μεγάλοι οργανισμοί, υπερβολικά μεγάλοι, και από τότε που δημιουργήθηκε η Τραπεζική Ένωση, το 1 τρίτο των τραπεζών εξαφανίστηκε. Έχουν γίνει τεράστιες συγχωνεύσει και μια συγκέντρωση εξαιρετικά ανησυχητική. Υπάρχει ε, έμεση δημόσια εγγύηση που προκύπτει από την κλίμακα και μόνο αυτών των δομών και αυτό δεν έχει λυθεί. Επίσης, το θέμα της εξυγίανση μας επισημαίνει πόσο σύνθετη είναι η κατάσταση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της Πορτογαλίας είναι σαφές ότι θα συνεχίσει αυτό να σημαίνει ότι τα, ε, το δημόσιο χρήμα θα, συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Στην τράπεζα Espírito Santo θα εξακολουθήσει η χώρα να πληρώνει 700 εκατομμύρια ευρώ υπό την έννοια, υπό τη μορφή εγγυήσεων που δόθηκαν στην περίοδο της εξυγένσης της τράπεζας. Και το ταμείο δεν είναι αρκετά αξιόπιστο. Άρα το θέμα πόρο απέχει από το να θεωρείται λήξαν. Ακούμε στοιχεία ότι δηλαδή οι μετοχές των τραπεζών είναι πολύ ισχυρότερε από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά έχουμε αύξηση κεφαλαίου λόγω της Βασιλείας 3. Και τα μοντέλα της αξιολόγησης της ε, ε, αξιολόγησης του ενεργητικού γίνονται από τις ίδιες τις τράπεζες, ε, εφαρμόζονται από τις τράπεζες. Πολύ απέχουμε από μια κατάσταση που θα μας δημιουργούσε αίσθημα εμπιστοσύνη για την πόσο, για το πόσο ισχυρό είναι το τραπεζικό σύστημα. Έχουμε πολλές αρνητικές πλευρές εδώ και γι' αυτό ακριβώς ανησυχώ. Όταν θα εμφανιστεί η επόμενη οικονομική κρίση, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα για, ε, στον τομέα της ευθύνη για μία ακόμα φορά. Ενδεχομένως θα δούμε ε, τις φοβερές συνθήκες που τόσο αρνητικά επηρεάζουν τη ζωή των Ευρωπαίων. Ο Μάρκο Βάλλη, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την πρότασή του. Πιστεύω ότι σε διάφορα σημεία πρέπει να τροποποιηθεί, διότι είναι διαφορετική η πολιτική μας τοποθέτηση. Θα υποβάλουμε διάφορες προτάσεις όπως γνωρίζετε. Η Τραπεζική Ένωση έχει διάφορα τμήματα και όσον αφορά την εποπτεία βλέπουμε διάφορα κρίσιμα σημεία όπου εκεί έχουμε συγκεντρώσει πολύ την προσοχή μας επί των πιστώσεων και στο κομμάτι των πιστώσεων που τελεί υποπίεση και λίγο στο χρηματοπιστωτικό κομμάτι δηλαδή τα στοιχεία ενεργητικού δευτέρου και τρίτου επίπεδου, στο οποίο έχουν αμειχθεί οι τράπεζε Γαλλία, Γερμανία και των βορείων χωρών, ε, αντιμετωπίζουν πολλού κινδύνου. και το είδαμε από τι δοκιμέ αντοχή που έγιναν φέτος ε, και ίσω να παρασυρώμεθα και να μην βλέπουμε τα σοβαρά προβλήματα και να δημιουργούν προβλήματα εκεί που δεν χρειαζόταν να δημιουργηθούν κι άλλα. Οι προτάσεις του εισηγητή να εισαγάγουμε ε, τα κρατικά χρέη. Ίσως πρέπει να δούμε τι γίνεται, τι βάρος θα έχουν στην εξολόγηση των τραπεζών για τον κίνδυνο. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο για τα τραπεζικά συστήματα και ενδεχόμενο οικονομικό κοινωνικό αντίκτυπο και σε όλη την ΩΝΕ. Ε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό πλευράς πολιτικής. Πρέπει να σταθμίσουμε με προσοχή αυτά που προτείνονται εμείς που ασκούμε πολιτική. Κυρίως εμείς ε, που ασχολούμαστε με το θέμα όσον αφορά την πρόταση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια χρειάζεται μια προσέγγιση για να τα αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε κάποιες χώρες όπως τη χώρα μου καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από τον τραπεζικό τομέα. Το θέμα είναι να μην δημιουργήσουμε πολλέ εντάσει και πίεση σε αυτή την κατεύθυνση. Διότι αν πολύ γρήγορα ή άμεσα με αυτόματου μηχανισμού αντιπιθυθούν αυτά τα μη ξυπηρεμούμενα χρέη, ίσω οδηγήσουν σε τραπεζικέ ε, κρίσεις πολύ βαθιές, που μετά θα την πληρώσουν οι πολίτες με του μηχανισμού εξυγίανση. Δεν είναι πάντα αυτόματη η λύση, αλλά δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Πριν τα εφαρμόσουμε αυτά, προτείνω εξαιρετική ευαισθησία και πολιτική ευθύνη από πλευρά αυτών που το προτείνουν και από φορείς όπως είναι η ΕΚΤ που αυτή θεσπίζει τους κανόνες, αλλά όχι μόνο η ΕΚΤ, αλλά εμείς μαζί με το Συμβούλιο. Δεν θέλουμε να εφαρμόσετε τόσο η πολιτική της ΕΚΤ, αλλά υποφάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που πρέπει να βρουν το σωστό πλαίσιο για την εφαρμογή των κανόνων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Όσον αφορά την έννοια της εξυγίανσης, Πρέπει να εξεταστούν οι ισχύοντε κανόνε, θα πρέπει να το συζητήσουμε με τον συνάδελφο ει βάθος και να εξετάσουμε και τις λεπτομέρειες. Η Ταπεζική Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί με επιμερισμό των κινδύνων και το περίφημο σχέδιο έχουμε με το Ταμείο Εγγυήσεων για τις καταθέσεις πρέπει αυτό να εξεταστεί το τάχιστο δυνατόν. Και αν ανεβάζουμε τον πύχη για τη μείωση των κινδύνων απομακρύνεται ο επιμερισμός των κινδύνων. Πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα, φτάσουμε στην Τραπεζική Ένωση. Και κάτι άλλο με το οποίο συμφωνούν πολλοί από τους συναδέλφους είναι και το άλλο. Το BSR, ο διαχωρισμός ο τραπεζικός είναι σημαντικό στοιχείο της Τραπεζικής Ένωσης. Το συζητήσαμε στην αρχή της θητείας, το συζητάμε πλέον αλλά ίσω να μπορούμε μέσω σωστή προσέγγιση να λύσουμε η ανδήποτε τραπεζική κρίση. Κύριε Λάγκε, δείξατε πολύ, είχατε μεγάλη ευέλιξη στον αυτό το χρόνο αγόρευση σήμερα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό είχατε. Ναι, και τώρα έχω, έχω μπόνους, λέει ο Λάγκε, θα το χρησιμοποιήσω. Θα το χρησιμοποιήσω για μένα, λέει ο πρόεδρο. όχι για τον κύριο Βάλλη. Ε, δεν έχουμε την ενέργεια, θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή εκ νέου. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Νομίζω ότι ε, μερικά από τα σημεία επί των οποίων διαφωνούν οι σκιώδεις είναι γνωστά από καιρό. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν τον μη ισοσκελισμένο προπολογισμό και την έλλειψη ε, παραγωγικότητας. Και βεβαίως αν αυτά δεν αλλάξουν δεν μπορούμε να φτιάξουμε το σύστημα. Το δεύτερο είναι ότι με κάθε σεβασμό, ε, συνάδελφε Βάλε, το κρατικό χρέος της Ιταλίας είναι ειδική περίπτωση. Ενδεχομένως να προσπαθήσουμε από κοινού να βρούμε μια λύση, αλλά δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο ότι υπάρχει δυνατότητα εξέβρεσης λύσης δηλαδή ότι ε, εσύ και εγώ μπορούμε να βρούμε τι θα γίνει. και να γλιτώσουμε. Να δούμε εδώ αν κάτι μπορεί να διορθωθεί. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το ανέφερα και αυτά στην έκθεσή μου. Όταν μιλάμε για τεράστια ζήτηση και αν πρόκειται να ξαναγράψουμε τους κανόνες από την αρχή, δεν νομίζω θα υπάρξει πλειοψηφία. Χαίρομαι που άκουσα τους ε, εισηγητές, εξω από τον Φίλιπ, αλλά αυτός θα επανέλθει αργότερα επί του θέματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χρονοδιά... Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι τροπολογίε μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τι 24 Οκτωβρίου, 19 Νοεμβρίου συζήτηση, 26 Νοεμβρίου ε, ψηφοφορία στην Ίκον και η, θα επιβεβαιωθεί η ψηφοφορία ε, στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Το επόμενο θέμα αφορά την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων και εισηγητή Σάντερ Λούς. Χαίρομαι που θα παρουσιάσω το θέμα, αλλά υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που θέλουν να ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη. Έχουμε εργότερα ψηφοφορία και Εν πάση περιπτώσει πρέπει να περιμένουμε άλλους συναδέλφους, οπότε στα γρήγορα να σε εξετάσουμε το θέμα, γιατί υπάρχει μία έκθεση στην ψηφοφορία, όχι δύο. Οπότε όλοι γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Η, η ίδρυση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται στην ε, ανοιχτή οικονομία αγορά. Το θέμα του ανταγωνισμού είναι βασική σημασία. Πάντοτε το στηρίζαμε εδώ και στηρίζαμε τις ε, προσπάθειες της Κομισιόν να εμποδίσει τη τρέβλες του ανταγωνισμού. Δεν είναι απόλυτα σαφές Ποιε είναι αυτέ οι στρεβλώσει του ανταγωνισμού, ποιοι είναι οι κανόνε και πώ πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη κλπ. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε έναν μηχανισμό που εισήχθη. Ο εξυγχρονισμός ε, ε, πρωτοβουλία της ε, κρατικής βοήθειας ξεκίνησε από την Κομισιόν με σκοπό να επικεντρωθεί στην εφαρμογή του δικαίου στις περιπτώσεις που επηρεάζουν περισσότερο τις εσωτερικές αγορές, η ζήτηση καλή συνεργασίας με τα κράτη-μέλη, την αποκέντρωση των ε, ευθυνών για την ε, εφαρμογή των μέτρων κρατικών ενισχύσεων, γιατί αυτό επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι οι εθνικές και περιφερειακές αρχές πολύ συχνά δεν εκτιμούν σωστά το θέμα ότι ε, τα κοινοτικά κονδύλια ε, αποκλείονται, εξαιρούνται από τα, ε, τους κανόνες της κρατικής, των κρατικών ενισχύσεων, είτε ότι ε, ε εμπίπτουν και αυτό σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα μπαίνουν στο άρθρο 107 εάν και μόνο εάν μπορεί η κρατική αρχή να τα ελέγξει. Και το θέμα είναι πώς μπορούμε να ε, μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη λειτουργία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε σχέση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και τώρα προτείνεται ε, μια αλλαγή ένας κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν θα μπορέσει η Κομισιόν να προτείνει γιατί ε, χρειάζονται το πεδίο του GPR για την χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Ταμεία. Άρα είναι τεχνικό το θέμα μάλλον. Προσωπικά στηρίζω την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτός και είναι και ο λόγος που προτείνω γιατί μιλάμε τώρα για την, τον πρόδρομο της ε, συζήτησης που θα ακολουθήσει, προτείνω να υπάρξει συζήτηση με βάση την απλουστευμένη διαδικασία. Δεν ξέρω αν ε, οι συνάδελφοι επιθυμούν κάτι άλλο. Ε, θα είμαι διατεθειμένος να δεχτώ και κάτι άλλο, αλλά λόγω και του φόρτου εργασίας της Επιτροπής μας, ενδεχομένως να περάσουμε με την απλουστευμένη διαδικασία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προτείνεις απλουστευμένη διαδικασία, έτσι δούμε αν, αν η θέση αυτή και των άλλων ομάδων. Το ΕΛΚ, ο Μάρκο, έχει το λόγο. Θα μιλήσω εκ μέρου του κυρίου, του συναδέλφου, της συναδέλφου πείτε. Κάινεν. Μου έδωσε μακρύ, μακροσκελή κατάλογο. Θα είμαι σύντομο. Εγκρίνουμε την προσέγγιση του εισηγητού σαν ΕΛΚ όσον αφορά το περιεχόμενο και την απλουστευμένη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ τη σύναψη αυτή. Οι σοσιαλιστές. Υπερβάνς. Εν ονόματι των σοσιαλιστών. Μιλώ εν ονόματι του συναδέλφου Μοργάνου που έπρεπε να μας εγκαταλείψει. Δεν μου έδωσε μακροσκελή κατάλογο να διαβάσω το μήνυμα ποιο είναι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή. Η πρόταση του συγητού προς τα προστευμένη διαδικασία για το θέμα της διάθρωσης μεταξύ ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μελλοντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων είναι μια καλή πρόταση. Την υποστηρίζουμε. Έξοχα. Ε, η Άλντε. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Όπως και ο Μάρκους Φέρμπερ και εγώ, σύντομα θα πω ότι εκτιμούμε τη δουλειά ε, του εισηγητού. Πιστεύω ότι κινούμεθα προς αποστευμένη διαδικασία και υποστηρίζουμε την προσέγγιση του όσον αφορά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Η πράσινη. Κανένα σχόλιο. Η Γκουε και εμείς υποστηρίζουμε την ε, συντομευμένη, την ταχεία αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ. Ωραία. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο εισηγητής θα παρουσιάσει την έκθεση που προς έγκριση στο Κοινοβούλιο θα υποβληθεί στην Ολομέρεια η έκθεση. Σύμφωνα με το άρθρο 50 ένα. Το τελευταίο σημείο. Ίδιοι πόροι. Α, ψηφοφορία, ψηφοφορία. Το συζητήσαμε αυτό πριν. Έχει επικαιροποιηθεί το κείμενο, αυτή είναι η εκδοχή μου. Κοιτάξτε, το φως με τυφλώνει και δεν σας βλέπω και πρέπει να σας βλέπω για την ψηφοφορία. Παρακαλώ, μπορούμε να κατεβάσουμε τα ρολά. Αν την καλοσύνη να καλυφθεί ο ήλιος τουλάχιστον. Σας παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη. Κάνουμε δοκιμή της ψηφοφορίας, άρχεται η ψηφοφορία. Μπορούμε να τελειώσουμε τη δοκιμή. Και μπορούμε Ας ξεκινήσουμε. Ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδοτήσεως Ραμόν Χερέγκα Τόντο για τους ιδίους πόρους. Τροπολογία 67 υπέρ. Κυρία Βίρνιχ, το μικρόφωνο σας. Θα ήθελα, λέει η κυρία Βίρνιχ, να πω κάτι. Λυπούμε για τον τρόπο που τον οποίο εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα. Οι συζητήσει περί συμβιβασμών έγινε χθε το βράδυ. Χθε το βράδυ, λοιπόν, δύο συμβαστικέ αναδιατυπώθηκαν. Μικρέ αλλαγέ τι κατανοώ. Αλλά συμβιβαστικέ E και G άλλαξαν σε σημαντικό βαθμό. Θα έπρεπε να είχαν συζητηθεί στη συνεδρίαση των σκιωδών και να μην είναι κάτι χαμένη ευκαιρία συμφωνία των σοσιαλιστών και του ΕΛΚ, να είναι αντικείμενο συμφωνία μεταξύ του χωρί να αμυχθούν οι άλλοι. Θα πρέπει οι δίβλοι επικοινωνία να παραμένουν ανοιχτοί. Ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το χαρτοφυλάκιο δεν ήταν καλό. Ανεπιτυχή ήταν η επικοινωνία τηλεφωνικά με την ομάδα του εισηγητού. Ο εισηγητή θέλει κάτι να πει. Παρακαλώ, ορίστε. Είσαι στην ομάδα ότι είχαμε μια συνεδρίαση των σκιωδών πριν από μια εβδομάδα και δυστυχώς ορισμένες πολιτικές ομάδες στις συμβαστικές μου έφτασαν χθες βράδυ. Δεν είχα λοιπόν τη δυνατότητα να οργανώσω άλλη συνεδρίαση σκιωδών γιατί ορισμένες πολιτικές ομάδες χρειάστηκε να κάνουν εσωτερικές συνεδριάσεις για να αποφασίσουν την ομάδα τους, ε, για να αποφασίσουν τη στάση τους έναντι των συμβασμών που είχα προσφέρει. Στη συνάδελφο της Άλτε ε, την παρακαλώ να καταλάβει ότι δεν είχα καμία άλλη δυνατότητα. Λυπάμαι, αλλά οι περισσότερες προτάσεις της συμπεριλαμβάνονται στο τελικό κείμενο. Σας ευχαριστώ. Ας ψηφίσουμε. Τροπολογία 67 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 70. Άρχεται η ψηφοφορία για την 70. Πέρας. Απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 και 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική α αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά η 16 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές υπέρ κατά κατά για τη 16 έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 83. Αντίστοιχο τμήμα 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83. Ε, 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76 και 77 και 78 υπέρ κατά αποχές Αδίκιο έχετε. 76-77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 78 υπέρ. Α, καταπίπτει. 80 λοιπόν. 80-81-82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 19 και 88 αποσύρονται, πάμε στην 87 και 89 μαζί, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, στην 90 και 92 πάμε μαζί, υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται, συμβιβαστική ΑΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 94 υπέρ κατά Έλεγχος για την 94. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 95 και 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική C υπέρ. C. Συμβιβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική E. Μάλλον τροπολογία 28 28 παρακαλώ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά Α, έλεγχος για 32, άρχεται η ψηφοφορία για την 32. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 20 με 19, μία ψήφος διαφορά. 33, υπέρ. Έλεγχος για την 33, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία, 20-20, άρα απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Η θέση της άλλης στην 36 κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά έλεγχος για τη 49. Άρχεται η ψηφοφορία. «49, πέρας, ισοψηφία 21-21, απορρίπτεται». Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. 49 ήταν αυτή που ψηφίσαμε. Και τώρα πάμε στην 50. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 52. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική. Όχι, όχι. 64. 64. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα Ψηφίζουμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω ετροποποίηθη με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 9 κατά, 3 αποχές, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Αν οι συνάδελφοι τη Επιτροπή Προπολογισμών, καλωσορίζουμε τον Ζαν Αχτουί, θέλετε να διακόψουμε ή μπορούμε να πάμε άμεσα στη ψηφοφορία. Πολύ καλά.